So, Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. με συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση της διάσκεψης των Πρόεδρων, που σήμερα είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη τους Ευρωβουλευτές σε σχέση με το ΕΛΚ θέλω να ευχαριστήσω θερμά που μας διέθεσαν την αίθουσά τους ως υποκατάστατο της Ολομέλειας για τη συνάντησή μας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε Ντόλ. Θα αισθάνεται στο σπίτι, στο σπίτι η κυρία Καγκελάριος Μέρκελ. Χαιρετίζω την Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας κυρία Άγγελα Μέρκελ που ήταν πρόθυμη να προσέλθει απόψε εδώ σε εμά die sich freundlicherweise bereit erklärt που ήταν πρόθυμη, δήλωσε ότι ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων με την διάσκεψη των Πρόεδρων μαζί μας. Για την διεξαγωγή της συνεδρίαση θέλω να προτείνω το εξής αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Μέρκερ μετά από μια εισαγωγική παρατήρηση δική μου θα παρέμβει εκείνη και θα μας προσφωνήσει. Μετά οι πρόεδροι των ομάδων και οι διορισμένοι από τα κόμματα, τι κοινοβουλευτικέ ομάδε, θα λάβουν τον λόγο θα ε, μιλήσουν για το χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους. Έχω μεγάλη παράκληση να τηρήσετε τον χρόνο σας ως αγορητές γιατί υπάρχουν ανηλμένες υποχρεώσεις για την συνέχεια και πρέπει να τηρήσω και την υποχρέωσή μου που έχω στο Λονδίνο αμέσως μετά στη συνέχεια. Κυρία Μέρκερ, είδατε εσείς ότι δεν βρισκόμαστε στην Ολομέλεια, ούτε έχουμε, καθόμαστε με την κατηγορία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πράγμα το οποίο στην αριστερή υπήρξε μεγαλύτερο χειροκρότημα όταν προσήλθατε. Ήταν αυτό προς έκπληξή μας, αλλά είναι προάγγελος αυτό για τα επόμενα που θα ακολουθήσουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Μέρκελ θα προσφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τη μορφή της ανοιχτής διάσκεψης των Προέδρων. Είμαι ευγνώμων. Αυτή την ημερομηνία πριν από αρκετό χρονικό διάστημα την είχαμε κανονίσει. Θα έπρεπε να είναι μια προσφώνηση ένας λόγος στην Ολομέλεια. Για τεχνικούς λόγους σήμερα δεν είναι αυτό εφικτό. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Έχω όμω την εντύπωση ότι έχει χαρακτήρα Ολομέλειας, αίθουσας Ολομέλειας αυτή η αίθουσα εδώ. Αυτό το μήνα θα έχουμε ένα έκτακτο συμβούλιο και από πλευράς ε, ε, καγκελαρίου για τις ε, διαβουλεύσεις για το μεσοπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε έντονα προπαρασκευάσει αυτή τη φάση. Γνωρίζετε τη, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επί της ουσίας και από πλευρά των δημοσιονομικών προτάσεων που έχει υποβάλει η Ευρωβουλή. Θέλω να επισημάνω ότι η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για την έκθεση των συναδέλφων Μπέγκε και Κάλφιν είναι η θέση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την μεσοπρό... τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό με πλειοψηφία άνω των 500 ψήφων και εγκρίθηκε από όλε τι κοινοβουλευτικές ομάδε. Είναι μια πλειοψηφία που καταδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει απόλυτα αυτή την απόφαση και όχι μόνο με μια μαχητική πλειοψηφία αλλά με μια ευρύτατη πλειοψηφία. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου στην έναρξη αυτής της συνεδρίασης να επισημάνω και να πω ότι κάθε που θέλει την επιτυχία της Ευρώπης πρέπει να είναι πρόθυμος για συμβιβασμούς. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι πρόθυμο να προβεί σε συμβιβασμούς. Έχουμε αφετηρίες, σημεία αφετηρίας που έχουμε καθορίσει, είναι σημεία αφετηρίας για τις διαπραγματεύσεις μας. Είμαστε πρόθυμοι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις στο τέλος να καταλήξουμε σε δίκαιους συμβιβασμούς. Λέω όμως ρητά, όποιος μας προαναγγέλει ότι υπάρχει μόνο μία θέση διαφορετικά αρνησή κυρία, βέτο, μην εκπλαγεί αν από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στην εκπροσώπηση στους αιρετούς εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών, υπάρξει και από αυτή την πλευρά αρνησή κυρία. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι πρόθυμο για συμβιβασμούς, αλλά είναι και μαχητικό και έτοιμο να δώσει μάχη. Ναι, μπορείτε να χειροκροτήσετε με την ησυχία σας. Χαίρομαι πέρα από αυτό για το ότι εσείς βρίσκεστε ανάμεσά μας σήμερα για να αναφερθείτε και στην ε, θεμελιώδη συζήτηση που θα έχουμε για τους νέους προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελλοντικά για τη μελλοντική διαμόρφωση της ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Χαίρομαι που μπορώ να σας δώσω τον λόγο να μας προσφωνήσετε. Έχετε τον λόγο κυρία Καγκελάρια. Μάλιστα κύριε αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μάρτιν Σούλτσα, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που σήμερα μπορώ να σας προσφωνήσω και είναι η πρώτη ευκαιρία από την Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου το 2007 και πάλι να βρεθώ ενώπιον σας και να σας προσφωνήσω και με χαρά δράτω με τις ευκαιρίες αυτής ώστε να εκφράσω τις απόψεις μου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο κυρίως ε, για την, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, αλλά και σίγουρα συζήτηση μπορεί να γίνει αυτό στη συνέχεια. Σε δύο ημέρες, την 9η Νοεμβρίου, θα έχουμε την επέτειο της πτώσης ε, του τείχους του Βερολίνου για 23η φορά. Η 9η Νοεμβρίου 1989 ήταν μια πραγματικά ευτυχή συγκυρία, μια ευτυχή στιγμή και της γερμανικής αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας συνολικά. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας εποχής ελευθερίας, ενότητας και δημοκρατία στη Γερμανία και στο σύνολο της Ευρώπης. Εμείς οι Γερμανοί ποτέ δεν ξεχνάμε ότι η ευτυχής εξέλιξη της δικής μας χώρας δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ ότι αυτό το οφείλουμε και στις θαραλές προσπάθειες για την ελευθερία ακριβώς των ανατολικών γειτόνων μας. Εμείς οι Γερμανοί γνωρίζουμε ποια είναι η ευθύνη μας για ένα θετικό μέλλον στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτή τη συνειδητοποίηση η Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση ασκεί πολιτική φυσικά για τη χώρα μας στην Γερμανία αλλά και για την Ευρώπη. Σήμερα θα ήθελα ένα κύριο στοιχείο, ένα κίνητρο, κινητήρα της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να υπενθυμίσω, την ελευθερία. Ελευθερία που καθιστά εφικτή την ζωή σε ε, ένα πλαίσιο ειρήνης και ευημερίας. Ελευθερία σε όλες τις πτυχές, ελευθερία της έκφρασης, ελευθερία των μέσων, του τύπου, της θρησκευτικής πίστης, του συναθρίζεστε. Όλα αυτά πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει πολυμορφία και δεν υπάρχει ανεκτικότητα. Η ελευθερία ελευθερία είναι τα θεμέλια, το θεμέλιο για την ενωμένη και την αποφασισμένη στεναρή Ευρώπη. Και ακριβώς σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που σήμερα πρέπει να περάσει η Ευρώπη για να αντέξει και να επιβιώσει. Μπορεί το να μας δώσει δύναμη να μπορέσουμε μέσα από την ελευθερία να βγούμε ενισχυμένοι και να μπορέσουμε να ηγηθούμε. Διότι η δύναμη της ελευθερίας δίνει ακόμα το θάρρος για αλλαγές, για μεταβολές. Είναι ακριβώς το θάρρος για τις αλλαγές που τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι το έχουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον διεθνή ανταγωνισμό του 21ου αιώνα να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει. Στα ταξίδια μου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στην Ήπειρο της Ασίας, κατά τα τελευταία χρόνια πολλές ε, δυναμικές, ε, φιλόδοξες ε, και χώρες που έχουν μεγάλη προοπτική γνώρισα. Εκεί με ενδιαφέρον στρέφουν το βλέμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές με ρωτούν με κάποια, θα έλεγα, με κάποιους δισταγμούς και σκεπτικισμό το ευρωπαϊκό πείραμα θα μπορέσει να αντέξει αυτή την κρίση. Αυτό το ερώτημα καταδεικνύει με σαφήνεια ότι αυτή η σοβαρή ε, κρίση που ε, διανύουμε σήμερα πραγματικά δίνει, πρέπει να δώσει μια προοπτική για ε, να, δούμε προς τα που θα κινηθούμε. Έτσι λοιπόν αυτό, αυτοί, αυτοί οι δισταγμοί μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να τα καταφέρουμε. Γι' αυτόν τον λόγο <clears throat> δεν είναι μόνο για αυτόν τον λόγο μια μεγάλη τιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση που τιμήθηκε με το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης. Πολύ περισσότερο από την έγκριση των συνθήκων της Ρώμης πριν από 55 χρόνια είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτική σημασίας μήνυμα και σήμα που σηματοδοτεί προς τον κόσμο και σε εμά τις ε, Ευρω... τους Ευρωπαίους πολίτες, γυναίκες και άνδρες ε, πώς πρέπει να κινηθούμε. Ο Μάρτιν Σούλτς το βραβείο Νόμπελ αποκοινούμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα, λάβουν αυτό, θα παραλάβουν αυτό το βραβείο στο Όσλο. Και χαίρομαι γιατί έχω αποφασίσει όπως και συνάδελφοί μου να συμμετάσχουμε σε αυτή την τελετή. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε με αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε όλοι, όλοι εμείς από κοινού, οι 500 εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι γνωρίζουμε, εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε ενωμένοι για την ευτυχία μας. Το βραβείο Νόμπελ μας δίνει ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό και να καταβάλουμε προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Είναι μια προειδοποίηση αυτό το βραβείο να θέσουμε πάλι στο επίκεντρο των πραγμάτων αυτά τα οποία είναι σημαντικά στη σημερινή συγκυρία κρίσης και όχι μόνο την υπερχρέωση, το μισθολογικό κόστος, ε, το ποσοστό ανάπτυξης, παρότι είναι όλα αυτά σημαντικά. Το πιο σημαντικό όμω είναι να αναγνωρίσουμε ότι το κοινό μας νόμισμα είναι κάτι παραπάνω από ένα κοινό νόμισμα. Είναι ένα σύμβολο για την επιτυχή ειρηνική και δημοκρατική ένωση της Ευρώπης. Ένα σύμβολο για την Ευρώπη της ελευθερίας, ε, της ευημερίας και της πρόοδου. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή για τίποτα άλλο δεν πρόκειται παρά για το ότι αυτή την ευτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την τύχη να την διασφαλίσουμε και να την, να την διατηρήσουμε και να την συνεχίσουμε για τα παιδιά μας. Γι' αυτό μας υποχρεώνει το βραβείο Νομπέλ να κάνουμε μια καλύτερη ένωση, μια Ευρώπη της σταθερότητας και της ε, δύναμης. Ο Μάρτιν Σούλτς είχε δίκιο όταν στον λόγο που προσφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκλεγής πρόεδρος είπε παράθεμα είτε θα χάσουμε όλοι μας είτε θα κερδίσουμε όλοι μας. Τέλος παραθέματος. Η κοινή μας ε, στάση, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι ότι θέλουμε και πρέπει από κοινού να κερδίσουμε όλοι. Αυτή είναι η θέση μας και από κοινού μπορούμε αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο της οικονομικής επιτυχίας και της κοινωνικής υπευθυνότητα να το, να το συνδέσουμε και να το διασφαλίσουμε, να το υπερασπιστούμε ακόμη παραπάνω. Από κοινού μπορούμε να το ενισχύσουμε περισσότερο από ό,τι ποτέ και από κοινού μπορούμε να έχουμε τη δύναμη της ελευθερίας και το θάρρος για τις αλλαγές. Πρώτες επιτυχίες αυτών των προσπαθειών για την υπέρβαση της κρίσης είναι ευδιάκριτες και στο επίπεδο των κρατών μελών και στην εκπόνηση νέων μέσων για την υπέρβαση υπέρβαση της κρίσης. Όμως φυσικά με τα όσα κερδίσαμε και επιτύχαμε δεν πρέπει να επαρκεστούμε. Πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν ώστε η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να ανακτηθεί. Γι' αυτό δεν πρέπει στα μισά του δρόμου να, να μείνουμε στάσιμοι. Θέλω να σας υποσχεθώ εδώ σήμερα. Η, Ευρώπη θα, η Γερμανία θα κάνει κάθε προσπάθεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον να μπορέσει να τηρήσει την ευθύνη της, την υπόσχεσή της για ελευθερία και ευημερία. Και βρίσκομαι εδώ και ζητώ και την δική σας υποστήριξη. Διότι πάλι εκείνες οι δυνάμεις ε, αυξάνονται που πιστεύουν ότι μπορούμε τώρα να εφησυχάσουμε και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν χρειάζεται να την ε, ανανεώσουμε διότι με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης ε, έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι λάθος λάθος εκβάθρον, Αντίθετα από το να εφησυχάσουμε πρέπει σε όλα τα επίπεδα βήμα προς βήμα να μεριμνήσουμε η δύναμη της Ευρώπης να ανακτηθεί. Ελευθερία, δυναμική, ευημερία που η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό μπορεί να προσφέρει. Η ανθεκτικότητα και οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω, στην παγκόσμια σκηνή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωζέ Μανουέ Μπαρόζο στον λόγο που εξεφώνησε για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου είπε παράθεμα πρέπει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να ολοκληρωθεί τέλος παραθέματος και πράγματι πρέπει τώρα να βρούμε την ορθή πορεία, ώστε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση διαρκέστερα να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να άρουμε, να μπορέσουμε να επανορθώσουμε τα σφάλματα που έγιναν. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Δεν μπορούμε απλά να πούμε σε σχέση με την αλλαγή μιας συνθήκης να υπαναχωρήσουμε ή να φοβηθούμε αν αυτό είναι αναγκαίο. Αυτή η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη και σε αυτό θεωρώ εσάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμμάχους, συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Για αυτή τη σημερινή κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο ή πρότυπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ξεχωριστό, μοναδικό δημιούργημα, ένα μοναδικό μόρφωμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε εκείνο για το οποίο η Ευρώπη δίκαια είναι ε, Πρέπει να βρούμε με επινοητικό εφάνταστο τρόπο κάτι και να δράσουμε όλοι για να βρεθούν νέε λύσει. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να προβούν σε μεταρρυθμίσει, διαρθωτικέ προσαρμογέ και αλλαγέ και μέτρα εξυγίανση διαρθωτικά και σταθεροποιητικά μέτρα, ώστε να κερδίσουμε την ανταγωνιστικότητά μα και ιδιαίτερα από την κρίση αυτή τα κράτη που πλήττονται απαιτούν πάρα πολλά από τους πολίτες. Και γνωρίζω πόσο υποφέρουν οι πολίτες σε αυτά τα κράτη που πλήττονται με αυτόν τον τρόπο. Το γνωρίζω αυτό, αλλά σε αυτή την δύσκολη συγκυρία μπορώ να δώσω ένα θετικό μήνυμα. Οι μεταρρυθμίσεις δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Οι κόποι δεν πήγαν στράφη, δεν ήταν μάταιοι. Και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Ελλάδα <coughs> είχαμε μια προσπάθεια σημαντική και το είδαμε, μειώθηκε το μισθολογικό κόστος. Και αυτός είναι ένα σημαντικός παράγοντας για να κερδίσουμε την ανταγωνιστικότητα. Ακόμα και τα ελλείμματα <coughs> όσον αφορά τον ισολογισμό μειώνονται και πρέπει να συνεχίσουμε με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, με την δημιουργία αυτής ε, της νέας ε, προσπάθειας διάσωσης, το ESM. Και τα δύο ανήκουν το ένα με το άλλο από κοινού και είναι σωστά και σημαντικά. Λοιπόν, η παγίωση η εξυγίανση και η ανάπτυξη πρέπει να συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Θέλω να το πω αυτό εδώ, διότι καμιά φορά αυτά τα δύο το ένα χρησιμοποιείται εναντίον του άλλου. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε μεγαλύτερη απασχόληση με βάση εξυ, ε, υγιείς προϋπολογισμούς. Αυτή είναι η προϋπόθεση για την, ε, τις μελλοντικές γενναίες, για να μην, η, να μην αφαιρεθούν οι ευκαιρίες από τη νέα γενιά η ανάπτυξη δεν είναι κάτι το οποίο πολιτικά μπορούμε εξάπαντος να καθορίσουμε. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους στην Ευρώπη που θα δράσουν ως επιχειρηματίες με το πνεύμα του επιχειρήν. Η επιχειρηματικότητα από την ελευθερία και την αναγκαία ελαστικότητα συναπαρτίζεται. Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού. Γι' αυτό στην Ευρώπη πρέπει να προβλεθούν μέτρα όπου η ανάπτυξη και η απασχόληση στα κράτη-μέλη θα ενισχυθεί. Και έχουμε ρητά και το δημοσιονομικό σύμφωνο, ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο συμπληρώνει παράλληλα την ε, πορεία αυτή ώστε να μπορέσουν στοχοθετημένα να χρησιμοποιούν τα δημόσια κονδύλια. Επειδή όμω μόνο με αυτό δεν μπορούν όλα να επιτευχθούν, πρέπει από την άλλη πλευρά να δημιουργηθούν νέε προποθέσει για νέα ανάπτυξη. Κυρίω με την ε, μετεξέλιξη τη ενιαία εσωτερική αγορά. Νομοθετικά μέτρα αυτού του συμφώνου πρέπει πολύ γοργά να υλοποιηθούν. Και έτσι θα απελευθερωθούν δυνάμει για την ανάπτυξη. Και αυτό θα είναι αποφασιστικό για το μέλλον μα. Το Συμβούλιο δεσμεύεται προ αυτή την προσπάθεια και είμαι πεισμένη ότι και το Κοινοβούλιο το ίδιο. Και φυσικά το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που σε δύο εβδομάδε θα αποφασιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σημαντικότατη προπόθεση ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε τα αναγκαία κίνητρα και την προώθηση για την ανάπτυξη. Και κάθε ευρώ, και αυτό πρέπει να είναι ο πύχη μα, ο γνώμονα μα, πρέπει να δίνει πρόσθετη αξία όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν φτάνει να δίνουμε κάποια χρήματα απλά. Πρέπει να υπάρχει στοχοθετημένη χρήση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και γι' αυτό οι πολιτικέ μα στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να επανεξεταστούν και να δράσουν αποτελεσματικά ώστε να μπορέσουμε τα αίτια τη κρίση να τα αντιμετωπίσουμε. Τα σφάλματα στην αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκή Νομισματική και Οικονομική Ένωση πρέπει να αναλυθούν για να μπορέσουμε να τα επανορθώσουμε. Είμαι πεισμένη, αν μπορέσουμε και τα δύο ταυτόχρονα να τα κάνουμε, μακροπρόθεσμα θα στεφθεί το εγχείρημα από επιτυχία. Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Με την συνθήκη του Μαστρίχ το 1992, πριν από 20 χρόνια, δημιουργήθηκε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Τότε <clears throat> οι αρμόδιοι της, ε, της Νομισματικής Ένωσης, εκείνοι που δημιούργησαν την Νομισματική Ένωση, δημιούργησαν παράλληλα με την Οικονομική Ένωση μια νομισματική ένωση που όμως ε, <clears throat> δεν βρήκε την επαρκή υποστήριξη. Έγινε μια νομισματική ένωση, η Οικονομική Ένωση παρέμεινε αδύναμη όμως. Με τα αποτελέσματα αυτής της ε, απόφασης που με την ε, εισαγωγή του ευρώ καταρχήν είχε αποκριβεί, όμως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, έχουμε να αγωνιστούμε για να επανορθώσουμε τα σφάλματα. Έτσι λοιπόν οι διαφορές ε, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν αντί να μειωθούν. Απλά και μόνο να δούμε την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους, αρκεί για να μας πείσει. Στα κράτη-μέλη <clears throat> επί χρόνια, παρόλα αυτά, ε, δημιουργήθηκαν ολόκληρα βουνά χρέους και μάλιστα είδαμε ότι σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν υπήρξαν κυρώσεις όπως θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί. Όλα αυτά δείχνουν με σαφήνεια. Τα προβλήματα τα οποία σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν έχουν τις ρίζες. Τα αίτια αυτά βρίσκονται πολύ πιο πίσω από την σημερινή ε, οικονομική συγκυρία, οικονομική κρίσης. Ακόμα έχουμε και την κρίση, ε, κρατική κρίση, τραπεζική κρίση, υπερχρέωση, υπερχρέωση του ιδιωτικού τομέα, ε, απουσία της ανταγωνιστικότητας. Σε κάποιες χώρες έχουμε πολλούς από αυτούς παράγοντες από κοινού που πρέπει να πούμε ότι υφίστανται από κοινού. Αν όλα τα κράτη-μέλη είχαν τηρήσει αυτές τις οριακές ε, τιμές που είχαν συμφωνηθεί για τα ελλείμματα, για τα χρέη και είχαν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, τότε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ποτέ, ακόμα και αν ήταν αδύναμη, δεν θα κατέληγε σε μια τέτοια κρίση. Έτσι όμως ε, το μείγμα από σφάλματα που έγιναν από την αρχή σχεδόν απέβησαν ολέθρια αυτά τα σφάλματα για την Ευρώπη και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μαθήματα από αυτή την κρίση που πρέπει να, συνα... να συναγάγουμε να μάθουμε, να μην επαναλάβουμε αυτά τα σφάλματα. Πρέπει να μεριμνήσουμε η Ευρώπη να ε, βγει ενισχυμένη από αυτή την κρίση. Όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν ότι οι παραλήψεις του παρελθόντος κατά την δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να αναλυθούν οι βάσεις και τα βάθρα πρέπει να ανανεωθούν. Και πέρα από αυτό πρέπει εθνικά στα κράτη-μέλη να δημιουργηθεί αξιοπιστία. Αξιοπιστία, επιτέλους να τηρηθούν όλα αυτά τα οποία υποχρεωθήκαμε να τηρήσουμε. Ένα παράδειγμα <clears throat> το ότι δεν το κάνουμε είναι ότι εμείς ως αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ή οι προηγούμενοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαμε συμφωνήσει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δίνουμε ε, το 3% του ΑΕΠΑ για την έρευνα και την ανάπτυξη έχουμε χώρες που δίνουν 0,7, άλλες που δίνουν 3,5%. Κανείς όμως δεν τήρησε πραγματικά αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει ουσιαστικά. Γι' αυτό για μένα, για το μέλλον, τέσσερα στοιχεία είναι σημαντικά ως άξονες. Πρώτον, μια ανανεωμένη οικονομική και νομισματική ένωση χρειάζεται περισσότερη οικονομική, δημοσιονομική πολιτική πρέπει να ε, βασίζεται σε λειτουργούσες και αποτελεσματικές αγορές ως πλαίσια. Πρέπει να καθορίσουμε τις συνθήκες και όρους πλαίσια για όλα αυτά και να εναρμονίσουμε τους, τις, ε, ε, τα όσα θα ισχύουν και να μεριμνήσουμε ότι θα μπορέσουν και οι διεθνείς αγορές να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει επίσης να έχουμε έναν ευρωπαϊκό αποτελεσματικό μηχανισμό για την εποπτεία των τραπεζών, ώστε οι συστημικοί κίνδυνοι όσον αφορά την οικονομική τάξη πραγμάτων να μπορέσουν έγκαιρα να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν επιβεβαιώσει ότι η ποιότητα είναι σημαντικότερη από την ταχύτητα. Γι' αυτό πρέπει τα περίπλοκα νομικά θέματα να αποσαφινιστούν πρώτα, διότι πρέπει να είναι μια τραπεζική εποπτεία αυθεντική που θα αξίζει αυτό τον τίτλο. Δεύτερον, μια ανανεωμένη οικονομική και νομισματική ένωση χρειάζεται κοινή, κοινό, κοινή εναρμονισμένη δημοσιονομική πολιτική. Με την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχία και με το δημοσιονομικό σύμφωνο κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Χαίρομαι για το ότι εντωμεταξύ 11 από τα 12 ε, κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει τελευταία η Γαλλία και η Εστονία. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα πηγαίναμε ακόμα πιο πέρα. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα, να έχουμε δικαιώματα πραγματική παρέμβαση έναντι των εθνικών προπολογισμών όπου τα όρια τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί, αν δεν τηρούνται, θα μπορούμε άμεσα να παρέμβουμε δημοσιονομικά για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Τρίτον, μια ανανεωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση χρειάζεται κοινή οικονομική πολιτική. Το βλέπουμε σήμερα με κάθε σαφήνεια. Απουσίαζε και απουσιάζει μια επαρκή δεσμευτική ε, προσπάθεια συντονισμού στο οικονομικό επίπεδο. Και έτσι δεν υπάρχουν δυνατότητες στην ε, Νομισματική Ένωση την αναγκαία κατεύθυνση της εθνικής δραστηριοποίησης ε, να την ακολουθούμε. Και θα πρέπει εδώ να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ώστε να επιβληθεί αυτό. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι. Ο παλαιότερος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, το 1989 στην έκθεση που υπέβαλε για τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης επεσήμανε ποια είναι η σπουδαιότητα και των δύο αυτών πυλώνων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Παράθεμα, το αναφέρω, μια νομισματική ένωση χωρίς επαρκή βαθμό <clears throat> οικονομικής σύγκλησης δεν θα μπορεί να υποστεί τις δοκιμασίες και έτσι μάλιστα θα είναι και επιβλαβής για την κοινότητα. Τέλος παραθέματος, Ζακ Ντελόρ 1989. Η κρίση κατέδειξε πόσο σωστή ήταν αυτή η ανάλυση του Ζακ Ντελόρ. Κατέδειξε ότι οι λανθασμένες εξελίξεις στα κράτη-μέλη πραγματικά την νομισματική ένωση μπόρεσαν να την οδηγήσουν στον να κλειδονιστεί και συνολικά αυτό απέβει επιζήμιο για το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι στον συντονισμό αυτό βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή στα σπάργανα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο κάναμε μια πρώτη συζήτηση για όλα αυτά και συμφωνούμε ότι σε εκείνα τα πεδία πολιτική που για τη λειτουργία τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα, στο μέλλον θα πρέπει επακριβέστερα και σε μεγαλύτερο βάθος και έγκαιρα να εξετάσουμε το τι γίνεται διότι η απώλεια της ανταγωνιστικότητας για ένα κράτος μέλος ταχύτατα θα γίνει πρόβλημα για όλα τα άλλα κράτη-μέλη ένας ε, πιο ενισχυμένος βαθμός οικονομικού συντονισμού, οικονομικού συντονισμού θα είναι αναγκαίος, ιδιαίτερα όπου θίγονται θέματα του πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών μελών, όπως για παράδειγμα πολιτικά πεδία όπως ε, την ε, αγορά, την κατάσταση της αγοράς ή την φορολογική πολιτική. Πρέπει εδώ φυσικά να σεβαστούμε τις διαδικασίες που ακολουθούνται και εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε όμως λύσεις που δημιουργούν μια σωστή ισορροπία μεταξύ της αναγκαίας επέμβασης στο ευρωπαϊκό επίπεδο και του επίπεδου που πρέπει να διασφαλιστεί για τη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών πεδίων ή τομέων στα κράτη-μέλη και των κοινοβουλίων τους. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να μπορέσουμε να αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε λάθος κινήσεις. Πρέπει επιτέλους να έχουμε μια ανταλλαγή μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου. Είμαι υπέρ μιας κλιμακούμενης, διαφοροποιούμενης διαδικασίας ε, που θα δίνει την δυνατότητα ενός πλαισίου ώστε τα κράτη-μέλη με την έγκριση των κοινοβουλίων τους να μπορούν να επιβάλλουν ε, μεταρρυθμίσεις που θα είναι δεσμευτικές ε, και στο ευρωπαϊκό επίπεδο να ακολουθούν παράλληλη πορεία. Μπορώ να φανταστώ ότι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις με στοχοθετημένη αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσουν κίνητρα ώστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να είμαστε αλληλέγγυοι. Εδώ έχουμε την ιδέα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζεται μια βιώσιμη αποτελεσματική νομική βάση και που θα αποφασίσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το, ε, του Δεκεμβρίου το τι θα πρέπει να γίνει και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Εγώ είμαι υπέρ του ότι τον Δεκέμβριο πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο δρομολόγιο, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα αποφασίσουμε με συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα που θα εμπεριέχει που τα επόμενα επόμενα δύο έως τρία χρόνια θα θέλουμε να εφαρμοστούν. Και συνοψίζοντα, θέλω για άλλη μια φορά να πω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κυρίω εταίρο μα. Εταίρο όλων μα. Δεν θέλουμε ούτε να διχάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση καθόλου. Ούτε θέλουμε να δημιουργηθεί κάτι κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Καθόλου. Εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρξει η αναγκαία αμφίδρομη δράση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε όπως είπε και ο Ζακ Ντελόρ προς μεγαλύτερο επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας μακροπρόθεσμα. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, η ευρωπαϊκή κρίση υπερχρέωσης είναι στον πυρήνα της και κρίση αξιοπιστίας. Αυτό βλέπει κανείς όταν μιλάμε επενδυτές εκτός Ευρώπης και η εμπιστοσύνη πρέπει πολύ προσεκτικά να ανακτηθεί για μια ανανέωση των θεμελίων της νομισματικής και οικονομικής ένωσης προς τους Ευρωπαίους πολίτες και προς όφελός τους που εσείς εκπροσωπείτε εδώ στην Ευρωβουλή συνολικά όλοι σας. Γι' αυτό βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Και όπως προανήγγυλα, ξέρω ποια είναι η ανησυχία για τον διχασμό ή κατακαιρματισμό της Ευρώπης, της Ευρωζώνης των 17 ή των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το μέλημα πρέπει να πιστικά να δράσουμε ώστε να υπάρξει εμβάθυνση της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης και απαραίτητο στοιχείο αυτό για, την, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον η ανανέωση της Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης για τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ πάντα θα προσκαλούμε να προσέλθουν γιατί είναι ένα, ένα θεσμικό όργανο ανοιχτού χαρακτήρα διότι όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ τουλάχιστον θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε η εμβάθυνση της ε, Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης να μην οδηγήσει σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων αλλά να οδηγήσει στην Ευρώπη της διπλής, διπλάσιας δύναμης. Και επιπλέον πιστεύω βαθιά ότι ο στόχος μιας Ευρώπης σταθερότητας και δύναμης μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν και αν τα κράτη-μέλη και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεργάζονται και θα συνεργαστούν από κοινού, όλοι και όλα τους. Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι υπάρχει ανησυχία της εθνικοποίησης του ευρωπαϊκού επίπεδου. Είμαι όμως πεισμένη ότι αν αυτά τα οποία έχουμε ενώπιόν μας καταφέρουμε να τα πετύχουμε με τον σωστό τρόπο, αν συναγάγουμε τα μάθη από αυτή την κρίση, τότε ακριβώς θα ζήσουμε και θα βιώσουμε και αυτό μάλιστα την τον εξευρωπαϊσμό του εθνικού επίπεδου. Αυτό θα βιώσουμε. Κάθε πολίτης θα βιώσει στη χώρα του ότι μόνο με την Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αν δραχθούμε αυτή τη ευκαιρία, αν κατανοήσουμε ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί από ότι τα επιμέρους έθνη της Ευρώπης, τότε θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημά μας. Και τα εθνικά κοινοβούλια όλο και περισσότερο θα επομίζονται τις ευθύνες τους για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών το ίδιο. Ο πρόεδρος ε, Φαν Ρόμποϊ σε έναν λόγο που εξεφώνησε <clears throat> προς αυτόν τον στόχο ήδη, παράθεμα αναφέρω, ανέφερε <clears throat> ότι είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτά, τα οποία έτσι τα χαρακτήρισε τα εθνικά κοινοβούλια. Η Ευρώπη λοιπόν είναι όλοι από κοινού. Η Ευρώπη είναι η εσωτερική πολιτική με άλλα λόγια. Γι' αυτό ένας ενδυναμωμένος, εμβαθμένος διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια πραγματικά θα βοηθούσε τους εθνικούς βουλευτές να επιτελέσουν καλύτερα το έργο τους για ένα καλύτερο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιτελέσουν αυτό το έργο και με καλύτερο τρόπο, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είμαι πεισμένη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε την Ευρώπη τη σταθερότητα και τη δύναμη. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευρω... Ε, δημοκρατική νομιμότητα, νομιμοποίηση και έλεγχο. Για μένα είναι αποφασιστική σημασία αυτή η νομιμοποίηση και αυτό ο έλεγχο να διεξάγονται σε εκείνο το επίπεδο που λαμβάνονται οι αποφάσει και εφαρμόζονται οι αποφάσει. Δηλαδή, αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού επίπεδου που θέλουμε να ενισχυθεί. Ε, τότε ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει φυσικά να ενισχυθεί εκείνο. όταν αφορώνται θέματα εθνικών αρμοδιοτήτων, φυσικά τα εθνικά κοινοβούλια θα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Και πρέπει ανοιχτά επιπλέον να συζητήσουμε για το πώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσεις που αφορούν μόνο την Ευρωζώνη στο μέλλον <clears throat> θα μπορούν να νομιμοποιούνται. Για παράδειγμα θα πρέπει να προβληματιστούμε, να στοχαστούμε. Μόνο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κρατών της Ευρωζώνης θα ψηφίζουν ή κάποιοι όπως υπήρξαν κάποιες υποθέσεις πιο πριν, θα πρέπει να δημιουργηθούν λέει, άλλα ε, κοινοβουλευτικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει εδώ να δρά. Ενισχυμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτέ τι αρχέ πρέπει να προσέξουμε και να σεβαστούμε. Αυτέ οι αρχέ είναι ο πυρήνα τη ανανεωμένη νέα Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, ε, νομισματική και οικονομική ένωση. Μόνο με νομιμοποίηση των κοινοβουλίων θα υπάρξει αυτή η δημοκρατική νομιμοποίηση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μια και σήμερα προσφωνώ και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη του, Υπενθυμίζω φυσικά το έτος 2007, το έτος της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Τότε, με αφορμή την 50η επέτειο της υπογραφής των συνθήκων της Ρώμης, εκφράσαμε την ε, πεποίθησή μας στην διακήρυξη του Βερολίνου. Ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Hans Pöttering, υπέγραψε το έγγραφο αυτό ε, εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υπογραφή της 25ης Μαρτίου 2007 μπορεί σε μια ιστορική ανασκόπηση να θεωρηθεί ως σημαντική προϋπόθεση μέσω διαπραγματεύσεων που οδήγησε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τότε πρόκειται για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Σήμερα θέλουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση να εμβαθύνουμε, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθεί σε νέα σταθερότητα και δύναμη. Στη διακήρυξη του Βερολίνου το 2007 αναφέρθηκε παράθεμα. Η, η ιστορία απευθύνει μήνυμα και προειδοποίηση σε μας να δημιουργήσουμε τα θεμέλια για την τύχη και την ευτυχία των μελλοντικών γενεών. Γι' αυτό πρέπει η πολιτική διαμόρφωση της Ευρώπης να αποκτήσει σάρκα και οστά. Τέλος παραθέματος. Μόνο αν γίνει αυτό θα μπορέσουμε να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων έναντι της ιστορικής μας ευθύνης. Στην αρχή του λόγου που, σας, ε, που ξεκίνησα να σας προσφωνώ, ρώτησα θα μπορέσει η Ευρώπη να αντέξει τη δοκιμασία αυτής της κρίσης. Ε, θα σας πω ποια είναι η απάντηση και τι θέλω να απαντήσω εγώ. Ω, ως ε, επιστήμον μπορώ να πω ότι με τα πειράματα γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στη φάση που πέρασε ενός πειράματος βγαίνει από αυτό το πείραμα και πρέπει να μπορέσουμε πραγματικά να ε, στέψ, στέψει με επιτυχία το εγχείρημά της, με σταθερότητα, με ε, δύναμη και με δυνατότητα ανάπτυξης ως ε, καγκελάριος μπορώ να πω ναι, θα συνεχίσουμε την επιτυχία αυτή, την ιστορική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχιστεί αυτή η επιτυχία και η Γερμανία θα συνεισφέρει προς αυτή την επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι επιτυχής μόνο αν έχει τη δύναμη που δίνει η ελευθερία ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν θάρρος και φάνταστο τρόπο δράσης. Γνωρίζουμε, ενωμένοι και αποφασισμένοι είμαστε πάντα πιο δυνατοί ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να μεριμνήσουμε για την ειρήνη, την ελευθερία και την ε, ευημερία. Να είμαστε πρότυπο ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τις άλλες υπήρους και άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας και τίποτα λιγότερο. Πιστεύω στο ευρωπαϊκό κοινό μας μέλλον, ενωμένοι για αυτή την τύχη και ευτυχία μας. United for the better, ενωμένοι για το καλύτερο. Unis pour le meilleur. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μέρκελ. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Θα δώσω πρώτα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για 7 λεπτά το λόγο, ο κύριος Ζωζεφ Ντόλ. Έξι. Α, εγώ ήθελα να είμαι γενναιόδωρος, αλλά ο Ζωζεφ θα μιλήσει έξι λεπτά μόνο. Αγαπητέ Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Μάρτιν Σούλτ, αγαπητή Καγκελάρια της Γερμανίας κυρία Μέρκελ, αγαπητοί συνάδελφοι, τιμή και ευχαρίστησή μας να σας έχουμε μαζί μας, Καγκελάριε αποφασιστική στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης. Εδώ και 60 χρόνια έχουμε ειρήνη, εφημερία και το βραβείο Νόμπελ που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα το τόνισε, το υπογράμισε, το είπατε κι εσείς. Ωστόσο βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα αφανούμε ικανοί να ξαναδώσουμε όθηση στην Ευρώπη στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας της ειρήνης και της εφημερίας Η συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μια εικόνα της επιλογής επιλογής που πρέπει να κάνουμε. Για μας στο ΕΛΚ ζήτημα δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά ζητήματα. Εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα. Το ζήτημα είναι πω θα στηρίξουμε ένα σχέδιο που να εγγυηθεί την ευημερία μας και το μέλλον μα και κυρίω θα στηρίξει την καινούργια γενιά. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι απαραίτητος για την υπέρβαση της κρίσης, ασφαλώς. Υπενθυμίζω ότι 90% του προϋπολογισμού της Ευρώπης που πάει στις επενδύσεις ε, όχι μόνο επιστρέφει στα κράτη-μέλη, αλλά χάρη σε αυτό η δράση του ως μοχλό φέρνει καινούριε επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σχέδιο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πολύ τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που από τη μία πλευρά μας υποστηρίζει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020, από την άλλη μας ζητά περισσότερες δεσμεύσεις, αλλά ταυτόχρονα μας περικόπτει τις δαπάνες. Χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται συνοχή, συνεκτικότητα. Δηλαδή, χρειάζεται ένας προϋπολογισμός στο ύψος των φιλοδοξιών μας, φυσικά προσαρμοσμένος στις δύσκολες στιγμές που διερχόμαστε. Χρειαζόμαστε επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην καινοτομία. Είναι ισχυρή μοχλή ανάπτυξης αυτή οι τρει μοχλοί. Δημιουργούν θέσεις τη εργασία σε όλη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι έχει έρθει ο καιρός να γίνει ένας, μια συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Χρειαζόμαστε ίδιους πόρους για να εγγυηθούμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και για να διαιωνίσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης να ανακουφίσουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Χρειαζόμαστε καινούριες δημοσιονομικές δυνατότητες για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αλήθεια. Κάποιοι στο Συμβούλιο θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός πρέπει, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας καινούριος μίνι προϋπολογισμός. Τι πάει να πει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τον κύριο, τον κύριο προϋπολογισμό, πώς θα χρηματοδοτήσουμε ένα δευτερεύοντα προϋπολογισμό. Ε, η φτωχή η λογική μου του χωρικού δεν μου επιτρέπει να καταλάβω αυτό το επιχείρημα. Εγώ θα ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να το καταλάβω. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική και νομισματική συνοχή. Έχουμε την απάντηση γι' αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την νομοθεσία που ήδη έχουμε. Έχουμε το σύμφωνο, το οποίο πρέπει να επικυρωθεί και, να αποτελέ... και η εσωτερική ενιαία αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι ο κοινοτήριος μοχλός μας για την ανάπτυξη. Επίσης, έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν έχουμε ανάγκη για καινούριου θεσμούς. Το είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ούτε έναν ίδιο προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη. Ε, το κοινοβούλιο είναι που ανήκει στην Ευρωζώνη. Στο πλαίσιο της διαφανούς υπεύθυνη δημοκρατικής συζήτησης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι που πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα. Και πρέπει να πούμε όπως το λένε κι άλλοι ότι η Ευρώπη δεν έχει, ε, έχει 26 κράτη-μέλη αντί για 27. Όλοι μιλούν για ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Απαντώ εγώ σε όλους, σε διευθυντές, σε δικαστές μιας αλφα εθνικότητας, σε στελέχη. Ε, θα τους πω, προσοχή, είναι ένα ερώτημα που συχνά μου θέτουν. Όσο αφορά ε, για την ε, Βρετανική μη συστηματική προσέγγιση. Ε, δεν είναι ευρωπαϊκή. Βλέπω με πραγματισμό τη μεγάλη συμμαχία μεταξύ των Βρετανών σοσιαλιστών και συντηρητικών. Και του ρωτώ και σας ρωτώ αν είναι απαραίτητο το επόμενο Συμβούλιο να συγκληθεί όταν ένα κράτος θέλει και μπορεί να μπλοκάρει τα πάντα όπως το προβλέπουν τα νομοθετικά κείμενα. Ας εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα να προάγουμε τα άλλα θέματα που μας απασχολούν. Για πρώτη φορά ένα εθνικό κοινοβούλιο απαγορεύει κάθε διαπραγμάτευση στον αρχηγό της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν πρόοδο αυτό. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάνω στους συμβιβασμούς, πάνω στη δική μας μέθοδο, την κοινοτική μέθοδο και όχι σε ένα σύνολο κανόνων μιας ελάχιστης εσωτερικής ενιαίας αγοράς. Η Ευρώπη βασίστηκε στην αξία της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης πρέπει να σταματήσουμε να βγαίνουμε στις συνόδους κορυφής και να μιλούμε μόνο στον εθνικό τύπο για τις επιτυχίες μας, λες και είναι εθνικές επιτυχίες. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να προάγουμε το ευρωπαϊκό συμφέρον και σας ευχαριστώ που είχατε αυτό το θάρρος κυρία Καγκελάριε. Η εθνική κυριαρχία είναι ευρωπαϊκή στις μέρες μας επειδή τα 27 εθνικώς κυρίαρχα ε, κράτη ε, δεν είναι ικανά μόνα τους να λύσουν την κρίση, γι' αυτό θέλουμε μια ευρωπαϊκή Βρετανία, μια ευρωπαϊκή Γαλλία, μια ευρωπαϊκή Γερμανία, αλλά θέλουμε κυρίως 27 ευρωπαϊκά κράτη. Κυρίως θέλουμε μια ενωμένη Ευρώπη, ολοκληρωμένη, πολιτική Ευρώπη. Αυτό είναι το πραγματικό ευρωπαϊκό συμφέρον και στα γερμανικά. Κυρία Μέρκελ, την ευρωπαϊκή ιστορία τη ζήσατε επάνω σας, στον ίδιο σας τον εαυτό, με μεγάλη ένταση. Η ευρωπαϊκή ιστορία μας δείχνει πόσο σοβαρή υπόθεση είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Εμείς σας εμπιστευόμαστε ότι ε, την ευρωπαϊκή ενοποίηση θα συνεχίσετε να την συνδιαμορφώνετε με δραστήριο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Ντόλ. Καλό ήταν λοιπόν που σας έδωσα τα 7 λεπτά. Το πιο δυναμικό χειροκρότημα ήταν ε, του συναδέλφου Κονμπέντιτ κυρία Καγκελάριε, και αυτό είναι κάτι καινούριο. Ο κύριος Σβόμποντα ε, από τη, για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε κυρία Μέρκελ σας γνωρίζω, σας εκτιμώ ως άνθρωπο, εκτιμώ τις προσπάθειές σας για την Ευρώπη. Δεν θα σας εκπλήξει αν πω ότι η τωρινή γερμανική κυβέρνηση κάνει μια πολιτική που ε, είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Ξέρετε ότι το γερμανικό οικονομικό θαύμα στηρίζεται ακριβώς στην ε, ε, ύπαρξη της συνοχής στην Ευρώπη. Με την πολιτική σας όμως και με την υποστήριξη της Τρόικας ε, ζητάτε κάτι που δεν θα το ζητούσατε ποτέ για τη Γερμανία, την καταστροφή των κοινωνικών δικτύων. Πήγατε πρόσφατα στην Ελλάδα, κάπως αργά, αλλά πήγατε. Και είπατε εκεί ότι πρέπει να συμφωνήσετε με την Τρόικα. Να τα βρείτε. Ξέρετε όμως ότι η Τρόικα είναι δεστρόικα αφού καταστρέφει τα κοινωνικά δίκτυα που τα χρειάζεστε εσείς στη Γερμανία ακριβώς για την επιτυχία της ανταγωνιστικότητάς σας. Μιλήσατε για την ελευθερία, καγκελάριε. Τα εκατομμύρια των ανέργων, τι να την κάνουν την ελευθερία αυτή. Πρόσφατα έχουμε σήμερα πάλι έχουμε καινούρια νούμερα αυξημένης ανεργίας στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά και να μην τα βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στον αριθμό, των αυξανόμενων των ανέργων. Κυρία Καγκελάριε, είπατε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αλλά γιατί διστάσατε τόσο πολύ. Γιατί δηλαδή θα έπρεπε να ε, φάσει ο, ο πρόεδρος Ολάντ να μιλήσει για την Τραπεζική Ένωση. Αν δεν υπάρχει δεν θα μπορέσει ούτε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ισπανία για παράδειγμα. Την Ισπανία και την Ιρλανδία δεν πρέπει να τις βοηθήσουμε. Πρέπει να τις αφήσουμε μόνες τους. Όχι. Πρέπει να βοηθήσουμε. Μιλήσατε κυρία Καγελάρη για την κρίση του χρέους να διορθώσω κάτι στην Ισπανία. Δεν επρόκειτο για κρίση δημοσίου χρέους. Δεν ήταν αυτή η ρίζα του κακού, αλλά το ιδιωτικό χρέος που οδήγησε σε τραπεζική κρίση και έπρεπε μετά να βοηθήσει το κράτος. Και σήμερα έχουμε ε, ε, διαφορές επιτοκίων που ούτε η Γερμανία, ούτε η Αυστρία, ούτε άλλες χώρες ε, μπορούν να τις αφήσουν να εξελίσσονται έτσι. Δεν μπορούμε να καθίσουμε και να επαναπαυόμαστε και να αφήνουμε αυτά, αυτές τις τεράστιες ψαλίδες στα επιτόκια ε, που δεν θα βοηθήσουν την Ελλάδα και άλλες χώρες να βγουν από την κρίση. Γιατί δεν ε, γιατί ε, δεν ε, χρησιμοποιείται το μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε και στη Γερμανία για το μηχανισμό απόσβεσης του χρέους. Αλλά δεν, μπορούμε, δεν, πρόκειται για την κοινοτικοποίηση των χρεών. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να παρουσιαστούμε μαζί στις κεφαλαίες μέσα από την κοινή μας παρουσία θα μπορούσαμε να μειώσουμε και τα επιτόκια, ακόμα και για εκείνες τις χώρες που ε, αλυσοδένονται από αυτές τις διαφορές των επιτοκίων που είναι απαράδεκτες με το σημερινό τους ύψος και με την τεράστια διαφορά. Μιλήσατε για τον Τελόρ, αλλά κυρία Καγκελάριε, εσείς αφηγείστε άλλη ευρωπαϊκή ιστορία από τον Ντελόρ που είπε πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις για παράδειγμα για τη συνοχή της Ευρώπης. Μιλήσατε για την ανάπτυξη, μιλήσατε για την, τις επενδύσεις στην έρευνα και την ε, εκπαίδευση. Μειώνονται όμως, μειώνονται μαζικά μάλιστα αυτές όταν επιβάλλεται πολιτική λιτότητα στις χώρες και δεν μπορούν πια να επενδύσουν στην έρευνα και την παιδεία. Αυτό είναι το απαράδεκτο. Κυρία Καγκελάριε, αφηγήστε άλλη Ευρωπα... ιστορία και από τον Τελόρ και από τον προκάτοχό σα ε, τον ε, τον Helmut Kohl. Ε, έχετε δικαίωμα να έχετε τη γνώμη σας, αλλά από την άλλη τα εκατομμύρια των ανέργων, η αυξανόμενη ενεργεία δεν σας ε, επιτρέπει να ε, κάνετε αυτή τη διαφοροποίηση. Ούτε μπορεί αυτή η εξέλιξη να μας αφήσει ψυχρούς και αδιάφορους. Ξαναγυρίζω στον προϋπολογισμό. Κυρία Καγκελάριε, έχετε μια στάση στον προϋπολογισμό που είναι πολύ πιο λογική από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Αλλά και εκεί είναι αποφασιστική σημασία να ξαναδούμε αυτό που είπατε το Horizon, 2020 και άλλα στοιχεία της έρευνας και της ανάπτυξης συνεχίσουν να περικόπτονται, ε, τότε ε, δεν θα πρέπει, τότε θα πρέπει να παρουσιαστείτε και να τονίσετε ότι δεν επιτρέπεται να περικόπτονται ε, κονδύλια τα οποία, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Τέλος, είστε φυσικός, μας το είπατε απόψε πάλι, Βεβαίω, είστε φυσικό, είστε υπέρ των πειραμάτων. Όταν όμω βλέπει κανεί ότι τα πειράματα δεν πετυχαίνουν, τότε θα πρέπει να τα σταματούμε και να βάζουμε μπρο κάτι άλλο. Όταν βλέπουμε ότι η ακραία πολιτική τη λιτότητα, δεν μιλώ για ε, εξοικονομήσει κονδυλίων. Όταν βλέπουμε ότι η λιτότητα δεν λειτουργεί, τότε θα πρέπει να επιχειρήσουμε μια πολιτική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, μια πολιτική επενδύσεων και απασχόληση. Γιατί θα πρέπει να μειώσουμε την ανεργία, ιδιαίτερα την ακραία ανεργία των νέων. Αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται να το δεχτούμε ε, εμείς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Καγκελάρη. Και τώρα εξ ονόματος των φιλελευθέρων ο κύριος Φερχόφστατ. Κυρία Μέρκελ, κυρία Καγκελάρη, ευχαριστώ καταρχήν για την παρέμβασή σας. Δεν το επαναλάβατε σήμερα το απόγευμα, αλλά πριν από λίγες μέρες είπατε ότι η κρίση θα μπορούσε να ε, περάσει σε πέντε χρόνια. Αυτό είπατε σε μια συνάντηση της Τσεντεού. Πρέπει να πω ότι είμαι αισιόδοξο εκφύσεως, αλλά ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι αμφιβάλλω γι' αυτό. Γιατί? Γιατί όλα τα μέτρα που εφαρμόζουμε σήμερα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα αν ταυτόχρονα δεν καταπιαστούμε με το πραγματικό αίτιο της κρίσης, ε, θεωρώ. Και το αίτιο το βαθύ της κρίσης είναι για μένα πολιτικό. Έχει βεβαίως και οικονομική επίπτωση. Βεβαίως υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσει, αλλά πρόκειται για πολιτική κυρίως κρίση. Και το, το, η ρίζα της κρίσης είναι η σημερινή έλλειψη ε, μιας κρατικής ε, οντότητας, μιας δημόσιας οντότητας ε, πίσω από τα νομίσματα. Δεν νομίζω ότι ένα νόμισμα μπορεί να υπάρχει χωρίς ε, κράτος να σας το αποδείξω με κάποια στοιχεία. Έχουμε 90% χρέος στην Ένωση σήμερα και πληρώνουμε κατά μέσον όρο επιτόκιο, ο κ. Σβόμποντα ανέφερε την Ιταλία και την Ισπανία, ο μέσος όρος για την Ευρωζώνη είναι σήμερα 5% με 90% χρέος. Και στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουν 103% χρέος, περισσότερο χρέος από ό,τι στην Ευρωζώνη και πληρώνουν επιτόκιο μικρότερο από 2%. Και Σήμερα οι Ιάπωνες είναι οι πρωταθλητές του χρέους με 226%, το διπλάσιο της Ιταλίας και το επιτόκιο που πληρώνουν είναι 1,5%, το χαμηλότερο στον κόσμο. Πώς γίνονται αυτά, πώς είναι δυνατά. Αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο χρέος να έχουν το, τα μικρότερα επιτόκια, η απάντηση και η εξήγηση είναι απλή. Υπάρχει κεντρικό κράτος στην Ιαπωνία ε, που στηρίζει το γεν και το δολάριο το στηρίζει ένας προϋπολογισμός του 24% του ΑΕΠ. Και, ε, να είμαστε ειλικρινείς, πίσω από το ευρώ δεν υπάρχει τίποτε αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ένας προϋπολογισμός 1% θεωρείται πολύ υψηλός από πολλούς συναδέλφους σας. Ίσως ε, κάτι που μπορείτε να κάνετε κυρία Μέρκελ είναι να αναφέρετε τα νούμερα αυτά Ίσως ε, ο κύριος, ε, στον κύριο Κάμερον ε, ίσως θα μπορούσατε να αναφέρετε τα στοιχεία αυτά. Ε, ας δούμε τη σημερινή πραγματικότητα. Μην θεωρούμε πια ότι με ημίμετρα θα λύσουμε το πρόβλημα του ευρώ. Το ευρώ δεν είναι βιώσιμο και μπορεί να καταρρεύσει αν δεν δημιουργήσουμε γνήσιο ευρωπαϊκό κράτος με όλα τα δομικά στοιχεία του, με όλα τα συστατικά του, όπως τα έχουν οι Αμερικανοί πριν από 200 χρόνια που τα ε, έθεσαν στη θέση τους. Ε, γνήσια ευρωπαϊκή ε, διακυβέρνηση ε, ευρωπαϊκή δημοκρατία, γνήσιο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ε, γνήσιο ευρωπαϊκό ε, Υπουργείο Οικονομικών και αγορές τραπεζικές. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα που έθεσε ο κύριος Βόμποντα των υπερβολικά ψηλών επιτοκίων σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η επιλογή μας. Ή θα κάνουμε το βήμα προς την Ομοσπονδιακή Ευρώπη ή θα έχουμε πρόβλημα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, μια λέξη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να, ξέρουμε, πρέπει να ξέρετε ότι ε, τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για σας, την καγκελάριο της Γερμανίας. Αλλά αυτό που είπατε για την περίπτωση του κυρίου Μέρς ε, ήταν για μας απαράδεκτο. Η γνώμη του Κοινοβουλίου ε, δείχνει σεβασμό και είναι και σαφέστατη. Αυτό που αναμένουμε είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως εσείς θα αντιμετωπίζετε το γερμανικό Bundestag για τα ε, ε, εθνικά σας θέματα. Είναι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία το ίδιο νομιμοποιημένη όπως και η γερμανική. Äh, και τώρα η συνάδελφος Ρεμπέκα Χάρμς από την ομάδα των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για το ότι ήρθατε να συζητήσετε μαζί μας κυρία Καγκελάρια. Σας θυμόμαστε ως την Ευρωπαία πολιτικό που την συνθήκη της Λισαβόνας την κατέστησε οικία στους Ευρωπαίους. Και γι' αυτό ιδιαίτερα έχουμε κοινό συμφέρον μαζί σας για την λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Δημοκρατία που θέλουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί σας. Κατανόησα ότι θέλετε να στείλετε το μήνυμα ότι κανείς στην Γερμανία δεν ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα να διχάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις προτάσεις που έρχονται από τη Γερμανία όμως εγώ διαφορετικά τις κατανόησα και θα ήθελα να καταστήσω σαφές για σας ότι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι στο μέλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε όταν θα πρόκειται για την λήψη σκληρών αποφάσεων όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και Δημοσιονομική Ένωση, για παράδειγμα οι Πολωνοί συνάδελφοι <coughs> θα, εγκαταλείψουν, θα εγκαταλείπουν την αίθουσα πριν από την ψηφοφορία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος που γνωρίζει την ευρωπαϊκή ιστορία ότι πραγματικά βρίσκεται πίσω από την, ε, την ιδέα να δημιουργηθεί ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εδώ υπάρχει φόβος ότι αυτή η ιδέα συνδέεται με έναν ειδικό προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη, όπου κανείς δεν μπορεί σήμερα να πει από πού θα αντληθούν αυτά τα κονδύλια για ένα τέτοιο προϋπολογισμό. Αλλά ίσως μπορείτε αυτά να τα συζητήσετε με τον κύριο Κάμερον. Και για τα θέματα της ευρωπαϊκής ιστορίας το θεωρώ θετικό, το ότι υπενθυμίσατε την ε, ελευθερία και την δημοκρατία. Όμως πιστεύω ότι όπως εγώ γνώρισα και γνωρίζω την Ανατολική Ευρώπη και την Νοτιοανατολική Ευρώπη ότι η υπόσχεση για καλύτερη ζωή και δικαιοσύνη ήταν ένα κίνητρο για τα μεγάλα κινήματα που ακριβώς ε, στην Ανατολική Ευρώπη σημειώθηκαν και δημιουργήθηκαν. Και αν δούμε το αποτέλεσμα της πολιτικής διαχείρισης της κρίσης και της κρίσης της πολιτικής, τότε δεν μπορώ να αναγνωρίσω ότι ο στόχος της δικαιοσύνης με το σωστό τρόπο ακολουθήθηκε και ακολουθείται. Το βλέπω πραγματικά πάρα πολύ αρνητικό το ότι έχουν φόβο οι πολίτες ε, στην Ευρώπη για το μέλλον τους. Η Ελλάδα είναι ένα μέρος της Ευρώπης όπου μπορεί κανείς να δει εκεί προς τα που μπορεί να οδηγήσει μια μονομερής, μια μονόπλευρη οικονομική πολιτική. Και για το ότι αναφέρεται ότι κάποιοι είναι κατά των εξοικονομήσεων, αυτό το οποίο είμαστε εναντίον εμείς, του οποίου είμαστε εναντίον, είναι η μονόπλευρη αυτή πολιτική. Και μπορεί κανείς να μετρήσει πάρα πολύ, πολλές φορές ε, που προσπαθήσαμε να συνεννοηθούμε με το Συμβούλιο το αποτέλεσμα των συναντήσεων του Συμβουλίου ήταν ε, από πλευρά των σοφών τώρα θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Πήγαν όμως χειρότερα και πάνε χειρότερα και βρισκόμαστε σε μια σπυροειδή εξέλιξη που επιδεινώνει τα πράγματα. Παρεξέκλειναν τα κράτη της Ευρώπης ε, αναμεταξύ τους και μεταξύ από το Διεθνές ε, Νομισματικό Ταμείο προαναγγέλλεται ότι αυτό αυτός ο φαύλος κύκλος οξύνεται και θα οξυνθεί αυτός ο φαύλος κύκλος που ξεκινά με την πολιτική λιτότητα και καταλήγει στην πολιτική ύφεση οξύνεται. Έχουμε την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλα κράτη που οδεύουν αυτή την ολέθρια πορεία. Και πιστεύω ότι εσείς ως φυσικός που αναλύετε τα πράγματα και τα γεγονότα θα πρέπει αυτά να τα λάβετε υπόψη. Η Γερμανία πρέπει να ξεπεράσει αυτή τη μονοβαρή, μονόδρομη πολιτική και να ξεκινήσει μια συζήτηση για νέα μέσα τα οποία κατ' Επιγόντως χρειαζόμαστε. Όχι μόνο για να σταθεροποιηθεί το ευρώ, αλλά για να μπορέσει να παραμείνει ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και τώρα, εξ ονόματος των ε, Ευρωπαίων ε, Συντηρητικών, Ευχαριστώ πολύ κυρία Καγκελάριε Έκανα μαθήματα, γερμανικών με τους συναδέλφους. Ως περιστασιακός αναγνώστης του Der Spiegel, ας ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν ε, δίνεται και μεγάλη σημασία σε αυτά που σας λένε σήμερα. Ε, υπάρχει επιχειρηματικό πνεύμα στη Γερμανία. Ε, υπάρχει διάθεση αλληλεγγύης. Αν υπήρχαν νομίζω ότι θα συναντιόμασταν εδώ υπό διαφορετικές συνθήκες και έχουμε μεγάλη συμπάθεια προς τους Γερμανούς φορολογούμενους γιατί ποτέ δεν τους είπαν 50 χρόνια πριν ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο θα απαιτούσε από αυτούς να κάνουν τόσο μεγάλες θυσίες για να υποστηρίξουν και να διαιωνίσουν το ευρωπαϊκό νόμισμα. Αν ήμουν Γερμανός φορολογούμενος μάλλον θα συμφωνούσα με τους συναδέλφους όπως ο κ. Σουσούτορο και ο και θα ήμουν αντίθετο αντίθετο με το να χρησιμοποιείτε το γερμανικό χρήμα για τη στήριξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένο που οι ηγέτε ε, αυτών των ε, κομμάτων λένε τόσο διαφορετικά πράγματα εδώ από αυτά που λένε στην πατρίδα του. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και συμφωνώ ότι ο δημοσιονομικός συντηρητισμός είναι κοινός νους. Και αυτό μας το θύμισε η Μάργαρετ Θάτσερ, μια ε, γυναίκα που ήταν πολύ γεωμένη στη γη και που δεν ήθελε να παίζει με τα χρήματα άλλων ανθρώπων. Και αν τα χρήματά μου ε, χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη του ευρώ, τότε θα ήθελα να υπάρχουν πραγμα... μέτρα αυστηρά ε, έτσι ώστε να μην μπορέσουν να γίνουν κι άλλες δαπάνες και και να μην υπάρξουν ατασταλίες στις χώρες που έχουν ε, τύχη υποστήριξης. Έχουμε δει τι συμβαίνει στην Ελλάδα όταν η εθνική κυριαρχία παραδίδεται στην ε, γερμανική εθνική κυριαρχία. Όταν δεν μπορεί κάθε χώρα να ασχοληθεί με το οικονομικό της πεπρωμένο, τότε φυσικά η κατάσταση θα εκτροχιαστεί και θα, υπάρχουν κοινωνικές ταραχές οι κυβερνητικές διευθετήσεις της Ευρωζώνης, για τις οποίες μιλήσατε και θέλετε να οργανώσετε, θα πάρουν χρόνια και ακόμα και η Γερμανία νομίζω δεν έχει αρκετά χρήματα για να μας δώσει τον απαραίτητο χρόνο για την εφαρμογή τους. Είδε, το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος έχει, αποχαλ... έχει εκτροχιαστεί η κάθε χώρα διαπραγματεύεται τα δικά της επιτόκια. Είμαι σίγουρος ότι η δική μου χώρα θα θελήσει να επιστρέψουν κάποια δικαιώματα και αρμοδιότητες πίσω στα κράτη-μέλη. Ε, μιλάτε όλοι για την ολοκληρωμένη Ευρώπη, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν συμμερίζονται όλοι αυτό το όραμα. Καλό είναι λοιπόν να ακούγετε και να, να αφουγκράζεστε αυτούς ε, στους οποίους υπαγορεύετε τις επιλογές σας. Ε, νομίζω ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις ίδιες θεμελιώδεις ε, ε δυσκολίες που ανέκαθεν αντιμετώπιζε. Είτε θα μπορέσουν οι χώρες οι οποίες είναι σκλαβωμένες στο ευρωπαϊκό νόμισμα να απελευθερωθούν από τις αλεσίδες τους και να επιστρέψουν στο δικό τους ε, νόμισμα. Ε, δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει. Ε, ο καθηγητής Κάρκος Μέρκερ έκανε κάποια πρόταση η οποία φυσικά είναι γελία. Θα θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας αυτή την κρίση και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει, συλλογική, υπάρχει γενική έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Στο τέλος, ο δρόμος ο, ο λόγος των προβλημάτων μας είναι η έλλειψη της οικονομικής ανάπτυξης και απαιτείται γι' αυτό οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε όλη την Ευρώπη και ελπίζω ότι εσείς στη Γερμανία θα αρχίσετε να υλοποιείτε κάποιες από αυτές τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. E Για την ομάδα EFD, ο κύριος σας απόγευμα όλοι. Ε, έτσι λοιπόν θα διαπραγματευτείτε καγκελάριε με τον David Cameron για τον προϋπολογισμό ε, στα πλαίσια του ελεγκτικού συνεδρίου και της ε, διαδικασίας που προηγήθηκε. Ε, οι περισσότεροι ζητούν περικοπές και βεβαίως θα αντιμετωπίσετε και το, την οργή στην Βρετανία που θα αναρωτιούνται γιατί θα πρέπει να πληρώνουν 553 δι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οπωσδήποτε όμως ε, φαντάζομαι ότι θα κερδίσετε τη μάχη με τον κύριο ε, Κάμερον. Όμως ε, το πραγματικό θέμα είναι η θέση της Βρετανίας στην Ένωση γιατί τώρα φαίνεται ατέριαστη η Βρετανία σαν ένα τετράγωνο που πρέπει να περάσει μέσα από ένα κύκλο πρέπει να πω ότι ε, δεν έχει μείνει τίποτα για να πει ο Βρετανός Πρωθυπουργός και να πει κάτι ε, μας θεωρούν ότι ε, ε και δεν αφήνουμε ε, κανένα περιθώριο. Όμως ε, πιστεύω ότι τώρα έχουμε μια λιγότερη δημοκρατική Ευρώπη και δεν μπορούμε να σας ακολουθήσουμε στο ταξίδι σας αυτό. Είτε πρόκειται για εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, είτε πρόκειται για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή την τραπεζική έρωση. Ο Κάμερον πολλές φορές αναγκάζεται να πάρει μια θέση που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο από όχι. Γιατί τώρα, και τώρα το Labour Party, οι εργατικοί ε, αρχίζουν τώρα να είναι σκεπτικιστές και να ανθίστανται, ε, δεν ε, κάνουν αυτές τις συζητήσεις. Τώρα υπάρχει αυξανόμενη εχθρότητα προς την, το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, πολλές φορές κατηγορούνται οι αγορές για τα λάθη της Ευρωζώνης. Δεν θα ήταν καλύτερα αν πηγαίνατε στην Downing Street και λέγατε στον κύριο Κάμερον «Ακούσε να δεις, δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Ήρθε ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει το θάρρος να το πει ο ίδιος. Αν του το πείτε όμως εσείς, μπορεί να παίξετε κάποιο ρόλο. Τι άλλο να πω, αυτό μόνο προτείνω. Ε, προτείνω ε, να, γίνει ένα, να υπάρξει ένα φιλικό διαζύγιο το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε πολύ πιο καλές σχέσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Και τώρα από την Ενωμένη Αριστερά η κυρία Τσίμερο. Ναι, στην Ομοσπονδιακή Αριστερά. Ξέρω τώρα αν θα πρέπει να δώσω συνέχεια. Συνάδελφοι, τον λόγο έχει η κυρία Ευρωβουλευτής Τσίμερ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο τον κύριο Κάμερον θα πρέπει να τον λυπηθώ. Εκείνο θα λυπηθεί. Κυρία Καγκελάρια, σήμερα επανειλημμένα αναφερθήκατε στην ιστορία. Καλό αυτό. Σήμερα, για παράδειγμα, δεν είχαμε και την νίκη του Ομπάμα. Είχαμε και την 95η επέτειο της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Θα το θυμόσαστε αυτό από τα κοινά σχολικά προγράμματα που είχαμε στην Ανατολική Γερμανία, έτσι. Μάλιστα. Την Damen δεν ήξερα ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση προξενεί τέτοιο ενθουσιασμό. Κυρία Τσίμερ, έχετε τον λόγο. Αυτή την Οκτωβριανή Επανάσταση, για αυτόν τον λόγο ανέφερα, γιατί εσείς και εγώ, όπως και άλλοι, ζήσαμε τους ανέμους των αλλαγών το 89 και ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι σε καμιά στιγμή οι κοινωνικές ελευθερίες ε, δεν μπορούσαν να συνδεθούν και συνδυαστούν με τις ε, κοινωνικές ελευθερίες. Και γι' αυτό σας λέω με την πολιτική έναντι της Ελλάδας και άλλων χωρών της περιφέρειας της Ευρώπης, μια πολιτική λιτότητας η οποία βασίζεται το να οδηγήσει τους ανθρώπους στη φτώχεια και να χάσουν τα ε, θεμέλια της επιβίωσής τους και εκατοντάδες επιχειρήσεις ε, να χρεοκοπούν, δεν θα έχει μέλλον. Η λιτότητα σκοτώνει. Αυτό το είπαν και ευρωβουλευτές της δικής μου ομάδας ε, και στην Ολομέλεια επαρκώς. Και θέλω να αναφερθώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κοινωνικά δικαιώματα, ένα θεσμικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πρόσφατα δια, διαπίστωσε ότι τουλάχιστον δύο μέτρα του μνημονίου στην Ελλάδα παραβιάζουν την κοινωνική χάρτα και είναι παράνομα. Αφενός το αίτημα, η απέτηση, ο ελάχιστος μισθός ε, για απασχολούμενους ε, κάτω από 25 ετών ε, να μειωθεί και η παράταση σε σχέση με την προστασία για απολύσει να καταργηθεί. Και αυτά αφορούν αυτά τα μέτρα ιδιαίτερα όσον αφορά και την παράταση όσον αφορά τον χρόνο εργασίας Όλα αυτά είναι σημεία όπου σας απευθύνω κατεπίγουσα έκκληση να τερματίσετε αυτή την πολιτική επιτέλους. Όλα αυτά δεν έχουν καμία προοπτική να οδηγήσουν σε επιτυχία. Μισθολογικές μειώσεις. Δεν μπορεί αυτά να μας παρουσιάζεται ως απόδειξη ότι οι μεταρρυθμίσεις λέει στέφονται με επιτυχία. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν μπορούν αυτά να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ωφελεί η ανταγωνιστικότητα όταν καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές ζωή των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη δεδομένων των εξελίξεων. Και πρόσφατα ακόμα, και θέλω να το προσθέσω αυτό, πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα, είχαμε ένα συνώνυμο για την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το συνώνυμο ήταν ε, πολιτική συνοχής και διαρθρωτική πολιτική. Μπορώ να σας πω ότι η αλληλεγγύη που βρισκόταν στα θεμέλια αυτής της πολιτικής, δεδομένη στη συζήτηση για το, το, τα πολιετή ε, δημοσιονομικά πλαίσια, πραγματικά δεν τηρείται. Το αίτημά μα είναι όχι λιγότερα χρήματα, αλλά περισσότερα χρήματα για την πολιτική συνοχής για τα έργα που πρέπει να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει μεγαλύτερα κονδύλια να διατεθούν για την πολιτική συνοχή. Σταματήστε πια να λέτε ότι το, ε, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αποτελείται από κάτι παραπάνω από 1,0 τόσο της εκατό του ΑΕΠ. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική που θα βασίζεται σε άλλες αρχές. Προτού μου αφαιρέσει ο πρόεδρος τον λόγο, παρακαλώ να τα λάβετε όλα αυτά υπόψη. Θα ήθελα να μου πείτε, μέσα στο Συμβούλιο υπάρχει έστω και ένα κράτος μέλος που μπορεί να εξηγήσει και να πει ότι με τις περικοπές που προβλέπονται για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την πολιτική ανάπτυξη που είναι κατεσχήνη, έσχος για μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι για τα όσα συμβαίνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις χώρες. Και τώρα περικόπτουμε στην προστασία από θεομηνίες, καταστροφές, ιδιαίτερα για την πολιτική, για την ανάπτυξη. 7 δις ευρώ δεν είναι δυνατόν αυτά να τα δεχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνέσχος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σίμερ. Τώρα για τους μη εγγεγραμμένους, Σόζα Βάγνερ παρακαλώ. Κυρία Μέρκελ, κυρία Καγκελάρια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας στην Ευρωβουλή. Δεν ξεχάσατε και δεν θα έπρεπε να ξεχνάτε ότι αυτό το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ο οίκος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή. Και τώρα ερώτησή μου προς εμάς, κυρία Καγκελάρια. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σε σχέση με το... Ε, τα, όσα έχουν αποφασιστεί τα ε, θεωρεί αντισυνταγματικά. Διότι επειδή εσείς ε, την ισότητα ευκαιριών την παραβιάζετε όσον αφορά την ισότητα των πολιτικών κομμάτων. Θα ήθελα σε αυτό να αναφερθώ την ε, τοποθέτηση το, της ε, Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ε, και του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Σώσαν Βάγνερ. Κυρία Μέρκελ παρακαλώ για να απαντήσει. ich mich... Μάλιστα. Θα ήθελα και σε σχέση με τον πρόεδρο είναι απλούστερο μπορώ να, να ομιλήσω εγώ όπως αναφέρθηκε. Θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα του κυρίου Ζωζεφ Ντόρ αρκετά κοινά σημεία έχουμε, αλλά τέθηκε ερώτημα για τον προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη που διαδραμάτισε ένα ρόλο στις αναφορές προηγούμενα. Εγώ αυτό που επιθυμώ είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να είναι μια μέρα μέλη της Ευρωζώνης. Έτσι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχαμε πει ότι θα έπρεπε να περάσουν 15 20 χρόνια και να μην είναι όλα τα ε, κράτη-μέλη, κράτη τότε άλλα ερωτήματα θα έπρεπε να είχαμε απαντήσει τότε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τοποθετηθούμε σε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Αυτό σημαίνει ότι ένας βαθμός δεσμευτικότητας δεν επιτυγχάνεται για όλα τα κράτη-μέλη. Επειδή κάποια κράτη-μέλη θέλουν να έχουν περισσότερες ελευθερίες για λογαριασμό τους. Αλλά εκείνα τα οποία θέλουν και πρέπει να είναι σε ένα κοινό νόμισμα, πρέπει να είναι πρόθυμα να αναλάβουν ένα υψηλότερο βαθμό δεσμευτικότητα. Αν άλλοι θέλουν να προσθεθούν σε αυτή τη λέσχη, με τα χαρά, αλλά δεν μπορούμε να τα υποχρεώσουμε. Τώρα, πρέπει να διαφοροποιήσουμε αφενό τη δεσμευτικότητα. Αφετέρου, αναγνωρίζω πάρα πολύ καλά, πρέπει να πω, ότι κάποιες αρμοδιότητες σε χώρες ε, που ασχολούνται ιδιαίτερα σήμερα με τη δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν ε, πρόθεσμα. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων για να έχουμε την καταπολέμηση ανεργία των νέων, ε, πρέπει να έχουμε καλά καταρτισμένους και εκπαιδευμένου νέου. Η Ισπανία και η Πορτογαλία πρέπει να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Θα μας πούν όμω, θα μας απαντήσουν, δεν μπορούμε να το κάνουμε στο άμεσο μέλλον, δεν έχουμε χρήματα. Πρέπει να θεθεί το θέμα δεσμευτικότητα για την Ισπανία και Πορτογαλία. χωρίς όμως να αναφέρεται από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια, δεν έχω κάποια ελπίδα ότι όλα τα κράτη, 27 κράτη-μέλη, θα συναποφασίσουν να γίνει αυτό άμεσα. Όλοι γνωρίζουν στην Ευρώπη ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αλλά δεν θα υπάρχει προθυμία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τώρα γι' αυτό με ρημνώ για το ευρώ, διότι αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό. Και τώρα αυτή η δεσμευτικότητα θα πρέπει να ισχύει και να υφίσταται. Και αν όλα έτσι μπορούσαν να λειτουργήσουν, ότι όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ήταν κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πιο ενισχυμένο πλαίσιο για τα διαθροτικά ταμεία, ταμείο συνοχής και να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και δεσμευτικότητα για όλους. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για το ευρώ. Ούτε μήνες δεν μας δίνουν οι διεθνείς αγορές για να μην αναφερθώ σε χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να βιαστούμε και να ενεργήσουμε άμεσα. Δεύτερον, προς τον κύριο Σβόμποντα. Όλα τα άκουσα όσα είπατε και τα σημείωσα. Και πιστεύω και εγώ ότι συμφωνούμε, πρέπει να πω. 50% ανεργία των νέων σε κάποια κράτη-μέλη, όχι μόνο τρομακτικό είναι αυτό, αλλά ουσιαστικά είναι ανάξιο της Ευρώπης ως γεγονός. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να αλλάξει αυτή η τάξη πραγμάτων. Ανέλαβα την εξουσία, υπήρχαν στην Γερμανία πάνω από 5 εκατομμύρια άνεργοι τότε. Και ένας λόγος για τον οποίο ήρθα έχει σχέση με το ότι η κόκκινη-πράσινη κυβέρνηση έκανε μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία που δημιούργησε αλλαγές σε σχέση και με την ίδια τη βάση αυτών των κομμάτων ενώ από πλευράς αντιπολίτευσης ε, υποστηρίχθηκαν. και έτσι ανέλαβα εγώ την εξουσία συζητήσεις ε, για την ε, αξιοπρέπεια των ανθρώπων για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Κανένα κόμμα στην Γερμανία δεν έδρεψε θετικούς καρπούς ε, από αυτές τις ε, ε, μεταβολές. Πέρασαν πάνω από πέντε χρόνια, τώρα έχουμε τα θετικά αποτελέσματα. Μειώθηκαν οι άνεργοι, έχουμε μια καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση και τώρα αν δούμε την Ευρώπη και περάσουμε στην Ευρώπη και πούμε υπάρχει μόνο μια τυφλή πολιτική λιτότητας και να αυταπατώμαστε και να λέμε σε αυτά τα κράτη δεν χρειάζονται διαθροτικές αλλαγές, ε τότε αυτό είναι τρομερό λάθος έναντι και των ίδιων των συνδικαλιστών και των εργαζομένων της Ευρώπης. Λάθος αυτό, δεν είναι σωστό. Η Ελλάδα κατέληξε σε δυσκολίες όταν το έλλειμμα ήταν 15%. Κανένας δεν επέβαλε κάποιους περιορισμούς. Φτάσαμε στο έλλειμμα του 15% και αποφάσισαν τα διεθνή θεσμικά όργανα να μην δανείζουν πλέον στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η έναρξη της κρίσης και της κατάστασης. Και όταν τώρα λέμε ότι είναι πολύ αρνητική η κατάσταση της Ελλάδα, ναι, είναι πράγματι αρνητική, αλλά πρέπει να πούμε, δεν είναι εντάξει κάθε φορά να γίνεται απεργία όταν πρέπει να γίνει μια ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι καλό και δεν είναι εντάξει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να εισπράξει από τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς τα κόμιστρα τα οποία πρέπει να εισπραχθούν. Δεν είναι εντάξει όταν έχουμε ένα ε, σύστημα φορολογικό το οποίο δεν μπορεί να εισπράξει φόρους. Αν στην Ευρώπη δεν είμαστε σε θέση φιλικά, φιλικά να τα πούμε αυτά ο ένας τον άλλο και κάνουμε ότι αυτοί οι οποίοι τα λένε είναι αρίανοι, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Είμαστε 19% του παγκόσμιου πληθυσμού, 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ παράγουμε και 50% των κοινωνικών δαπανών έχουμε. Όποιος πιστεύει ότι όλα αυτά μπορούν να διατηρηθούν χωρίς ε, διαθροτικές αλλαγές, όποιος πιστεύει ότι με θολή αγορά εργασίας μπορούμε να προχωρήσουμε και με ανεργία των νέων δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και με την πείρα που έχουμε από την Γερμανία που είδαμε ότι είναι σωστή μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν έπρεπε να γίνει, τα δικά μας συνδικάτα στην Γερμανία και μέχρι σήμερα έχουν ε, ε, δισταγμούς και επιφυλάξεις για την αύξηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, τότε οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη να δράσουν υπεύθυνα για να πείσουν και να αλλάξουν τα πράγματα. Εκεί που πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη, εκεί όπου εφησύχασε, που δεν είδε τι συνέβαινε στις άλλες υπήρους και αλλού στον κόσμο, ε, ένα τεράστιο ποσοστό της οικονομικής ανάπτυξης διεξάγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κλείσουμε τα μάτια τότε δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, πραγματικά κύριε Φεχόφστατ λείπει η κρατική οντότητα αλλά αποτύχαμε σε σχέση με τη συνταγματική συνθήκη. Χάσαμε το δημοψήφισμα στη Γαλλία, χάσαμε το δημοψήφισμα στην Ολλανδία. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες της Ευρώπης να κινητοποιηθούν και να κινηθούν προ μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρώπης. Δεν μπορούμε όμως τα θετικά να τα πολέσουμε μαζί με τα αρνητικά που θέλουμε να ξεφορτωθούμε. Και δεν είναι δυνατόν αν θέλουμε να δράσουμε σωστά να αγνοήσουμε τις διαθωτικές αλλαγές που χρειαζόμαστε και τα θετικά. Τι συνέβη σε σχέση με την εισαγωγή του ευρώ. Παντού ήταν τα επιτόκια χαμηλά, όμως η ανταγωνιστικότητα κάποιων κρατών μελών επιδεινώθηκε. Και γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε τα κονδύλια μας, τα χρήματά μας να χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των πραγμάτων και της ευημερία. Και είμαι υπέρ του ότι κάποια μέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνει ένα είδους ευρωπαϊκή κυβέρνηση και το Συμβούλιο να γίνει ένα δεύτερο σώμα νομοθετικό στην Ευρώπη. Σήμερα όμως πρέπει πρώτα να διασώσουμε το ευρώ. Αυτό πρέπει να γίνει πρώτα. Να θέσουμε σωστά τα θεμέλια πρώτα. Να αφήσουμε λίγο χρόνο στους ανθρώπους για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και να πετύχουμε. Και σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Χάρμς, Ξέρετε και από τη Γερμανία, ας μιλήσουμε ειλικρινά, δεν ασκείται μονομερής πολιτική λιτότητας. Να σας πω κάτι, οι χώρες που έχουν ένα πρόγραμμα έχουν επιτυχίες σε σχέση με διαθροτικές μεταβολές. Έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι με τις ε, εξοικονομήσεις μέσα από την πολιτική λιτότητα. Παρότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια καλύτερη μεταρρύθμιση της αγοράς. Αυτή η προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα είναι αυτή που απαιτείται. Διαθωτικές αλλαγές. Δύο λόγια για τη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ θέλω μια ισχυρή Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω ξεκάθαρα. Είμαι Γερμανίδα. Η Μεγάλη Βρετανία μας βοήθησε να απελευθερωθούμε από τον εθνικό σοσιαλισμό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα μπορούσε να ανήκει η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρώπη. Και είναι καλό και για την ίδια τη Μεγάλη Βρετανία να ανήκει στην Ευρώπη. Σε ένα κόσμο 7 δισεκατομμυρίων να είναι μια χώρα μόνη τη δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό αυτό για τη Μεγάλη Βρετανία. Θα κάνω κάθε προσπάθεια η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι καλό εταίρο και γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Γι' αυτό θα πάω στο Λονδίνο. Και πραγματικά αυτή την υπέροχη νήσο θέλω να παρακαλέσω και να πω σε αυτό το νησί μπορείτε να είσαστε ευτυχισμένοι. Αλλά μόνοι σας δεν μπορεί να είσαστε ευτυχισμένοι. Είμαστε μια ισχυρή Ευρώπη 500 εκατομμυρίων πολιτών υπέρ της ελευθερίας της έκφραση, υπέρ τη ελευθερία τη δημοκρατία. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να είμαστε ισχυροί. Διαφορετικά δεν θα πετύχουμε. Ευχαριστώ. Για την κυρία Τσίμερ το εξή. Είπατε τόσο ωραία για το wind of change, τον άνεμο της αλλαγής το 89 που διήσε στις ελευθερίες. Αυτό που δεν είχε δει ο σοσιαλισμός ήταν ότι ε, οι κοινωνικές και οι προσωπικές ελευθερίες πάνε μαζί. Σωστό. Κάτι άλλο όμως ε, που παραγνώρισε ο σοσιαλισμός επίσης ήταν ότι δεν μπορούμε πάνω από τους ανθρώπους να κάνουμε οικονομία. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε μόνο σχεδιασμένη οικονομία, γιατί στερούμε τον κόσμο από την δημιουργικότητα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, σήμερα ε, δεν, υπάρχει, δεν είναι σωστός ο καταμερισμός που παραβλέπει τον επιχειρηματία, τον φορολογούμενο. Θα πρέπει οι φόροι να πληρώνονται, οι επιχειρηματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στην ε, ε, ε, σφαίρα του χρήματος. Θα πρέπει όμως όλοι και εσείς να κάνουμε τη δουλειά μας γι' αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι στη Γερμανία ε, να μην επικρίνουμε, να μην κάνουμε κριτική στις αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού μας Δικαστηρίου. Αυτές απλώς τις δεχόμαστε. Θα δούμε, το, το Γερμανικό Κοινοβούλιο θα συναγάγει κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να ε, επιχειρήσουμε κάτι το οποίο δεν θα μας οδηγήσει ε, σε επιτυχία, αλλά πάλι σε μια αποτυχία. Δεν ε, επικρίνουμε λοιπόν ε, και τις ε, αποφάσεις αυτές. Αυτή η απόφαση δεν ήταν σωστή και δεν αντικατοπτρίζει την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να το πει. Προτείνω τώρα... Α, κύριε Σόζα Βάγνερ, έχετε το λόγο. Κυρία ε, καγκελάριε, μου απαντήσατε διεξοδικά και σας ευχαριστώ πολύ. Μα εσείς είστε καταπληκτικός στην οικονομία του χρόνου σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Φαρατς. Είναι μια πολύ διαφορετική Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Οι 17 χώρες της Ευρωζώνης έχουν σαλπάρει στο δικό τους ε, ταξίδι και σε κάθε καινούργια πρόταση που έχετε υποβάλει, ο κύριος Κάμερον αναγκάστηκε να πει όχι. Τελικά θα βρεθούμε να είμαστε το κράτος στα χτωπούτα. Εσείς θα λαμβάνετε αποφάσεις για την ενιαία αγορά της οποίας είστε μέλος και, και, τα, και πάνω στα θέματα αυτά που θα έχουν συνέπειες στην Ευρωζώνη ε, είναι θέματα πάνω στα οποία εμείς δεν θα μπορούμε να ψηφίζουμε. Ειλικρινώς θα βρεθούμε σε μια εντελώς παράλογη θέση. Νομίζω ότι η Βρετανία είτε πρέπει να μπει πλήρω μέσα, είτε πρέπει να βγει πλήρω έξω. Ε, ίσως ο κύριος Κάμερο να συμφωνεί μαζί σας, αλλά ε, στα τελευταία ανάλυση ο, ο Βρετανικός λαός θέλει κάτι το εντελώς διαφορετικό. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίμερ, πολύ σύντομα, επί δύο σημείων, για την οικονομία. Η οικονομική πολιτική ως ε, βάση για την αναδιανομή και την εφαρμογή κοινωνικών δικαιωμάτων. Ναι σε αυτό, αλλά τα επόμενα 15-20 χρόνια στις πλέον θυγόμενες χώρες από την κρίση δεν θα είναι δυνατόν να οικοδομηθούν βιώσιμες οικονομικές βάσεις. Πείτε μου, με αυτή την πολιτική λιτότητα, ε, η, στρατηγική βιωσιμότητα της Ευρώπης πώς θα εφαρμοστεί ούτω ώστε να μπορούμε να αναπτυχθούμε σε πολλά επίπεδα. Επίσης, κάποια στιγμή μας είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικός εταίρος σας σε όλα τα θέματα καταπολέμησης της κρίσης. Γιατί τότε το δημοσιονομικό σύμφωνο δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε όταν είναι σαφές ότι σε δύο σημεία το σύμφωνο αυτό δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ουσιαστικά και τυπικά. Ε, δεν ε, αποφασίστηκαν ε, θέματα διεξαγωγής και εφαρμογής του συμφώνου από την Κομισιόν. Από τι θα συνοδεύεται όταν παραμερίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ε, την πρώτη πρώτου το δημοσιονομικό σύμφωνο θα τεθεί σε εφαρμογή, αλλά δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή την αντίφαση πώς θα τη λύσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλεναν. Καγκελάρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σίγουρα αναλωθήκαμε σε πολιτικές ρητορίες, ε, δεν αναφερθήκαμε στις, ε, στην οικονομική πραγματικότητα των χωρών. Κάποιοι ε, ανέφεραν ότι η Οκτωβρανή Επανάσταση, ο θάνατος 40 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι κάτι το οποίο πρέπει να πανηγυρίζουμε. Τέλος πάντων, κυρία Καγκελάρη, σας εύχομαι κάθε τύχη στη συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό μας απόψε. Φυσικά είμαστε μέλη των εθνών και μας ζητάτε να εφαρμόσουμε δημοσιονομική πεθαρχία κτλ. Σίγουρα ο κύριος Κάμερον μπορεί να, βασίζεται στην στήριξη των ε, ομοειδεατών του. Ε, κρίμα που το δικό σας κόμμα δεν σας στηρίζει πλήρως. Ε, θέλουν μάλιστα να ιδρύσουν και ένα μουσείο εδώ στις Βρυξέλλες. Ελπίζω να μπορέσετε να συνομιλήσετε μαζί τους και να πείτε ότι αυτά δεν είναι λογική επένδυση. Σε όλη την Ήπειρο, επιχειρηματίες, οικογένειες και πολίτες πρέπει να κερδίζουν όλο και λιγότερο. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει το ίδιο, να περικόψει τον προϋπολογισμό της. Δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προϋπολογισμό, αλλά καλύτερη χρήση του υφιστάμενου προϋπολογισμού και πιστεύω ότι ο κύριος Κάμερος θα, θα προωθήσει το θέμα των περικοπών του προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και το εργατικό κόμμα και η ομάδα του κύριου Σουόποτα θέλουν να περικοπεί ο προϋπολογισμός. Σε αυτό το περιβάλλον ζούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και να, αυξάνεται συνεχώς χρόνο με το χρόνο ο κοινοτικό προϋπολογισμός όταν επιβάλλεται λιτότητα σε τόσες χώρες και περικοπές σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες με τρόπο που είναι παντελώς μη αηφόρο είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Κάμερον θα κάνει τα δέοντα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμς έχει το λόγο. Να παρατηρήσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο το θεωρώ όχι ένα κράτος, αλλά ένα, μια χώρα που χρειάζεται πολύ εσωτερικές μεταρρυθμίσεις μετά την ε, ε βιομηχανοποίηση. Χαιρετισμούς ε, στους κυρίους Κάμερον και Μίλιμπαντα. Νομίζω ότι με την αντιευρωπαϊκή στάση τους δεν θα κρατήσουν σε υγιή τροχιά τη χώρα αυτή. Εγώ αύριο θα πάω στην Ελλάδα. Έχω ασχοληθεί με την ε, επικαιρότητα στη χώρα αυτή και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτούμε ότι με τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ε, έφτασε το τέλος. Ε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Ε, μείωσαν στο μισό μισθούς, συντάξεις, ε, πράγμα που θα ήταν απαράδεκτο στη Γερμανία οποιαδήποτε ιστορική στιγμή. Υπάρχουν όρια και στην πολιτική λιτότητα που εφαρμόστηκε στη Γερμανία. Τώρα η χώρα αυτή βρίσκεται στη χειρότερη οικονομική κρίση που θα οδηγήσει σε καταστροφή και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Κυρία Μέρκελ, αν η ε, Έλληνες δεν μπορούν να διατηρήσουν τη θέση τους κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες, δεν θα μπορέσουν ούτε οι άλλες χώρες να το καταφέρουν. Είναι πραγματικά ντροπή που η Γερμανία και κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες ακόμα πλούσιες χώρες πειραματίζονται πάνω στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σωστές διορθώσεις, τα διορθωτικά μέτρα γίνονται μόνο όταν η κρίση χτυπήσει τη δική τους την πόρτα. Ε, ακόμα ε, αντέχετε να το κάνετε αυτό, αλλά όχι για πολύ. Πρώτα η, η, πολιτική που λέει πρώτα μεταρρύθμιση στα κράτη-μέλη και μετά θα ακολουθήσουμε κι εμείς με περισσότερη οικονομική και νομισματική ένωση και πιο κοινέ αποφάσεις και περισσότερη κοινή ευθύνη, δεν αρκεί για, ε, αλλά θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η πολιτική αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι η πορεία που εκπροσωπείτε εσείς δεν δικαιολογείται πια. Ο κύριος, ε, ο κύριος Τρισέκε, ο κύριος ε, Ντράγκη είχαν αποφασίσει να ξεπεράσουν την ε, δυσφορία που υπάρχει τώρα θα μπορούσαν να κάνουν μια διαφορετική πολιτική αγορών και έτσι θα ερχόταν το τέλος αυτής της ε, κατάστασης με τον αποκλεισμό ε, που δημιουργείται από τις χώρες που ακόμα θεωρούνται ότι είναι οι χώρες που προσφέρουν. Ο κύριος Φερχόφστατ. Ναι, δεν νομίζω ότι διαφωνούμε για το μακροπρόθεσμο αλλά το θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων βημάτων. Λένε, λέτε ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε να υπάρχουν ε, ομοσπονδιακή διακυβέρνηση, ομοσπονδιακή ε, διακυβέρνηση των οικονομικών. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε τώρα όλα αυτά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώ η κρίση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στι μεταρρυθμίσει. Ένα παράδειγμα με τα επιτόκια. Τι γίνεται σήμερα. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι τα μισά μέτρα λιτότητα. Εγώ δεν είμαι κατά της λιτότητας στο νότο της Ευρώπης. Χρειάζεται για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αλλά τα μισά κέρδη από τη λιτότητα είναι για να πληρωθούν τα υψηλά επιτόκια των ομολογιούχων εκτός Ευρώπης. Ε, τα ε, χρήματα των Γερμανών φορολογουμένων πάνε για υψηλά επιτόκια που θα ωφελήσουν τους ομολογιούχους εκτός Ευρώπης. Αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχει ένας ευφυής τρόπος ε, επίλυσης. Προέρχεται από το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων, το Ζαχ Verständigen Rat, τους δικούς σας οικονομικούς συμβούλους που σας λένε κάντε ε, αμοιβαιοποίηση του χρέους όταν είναι πάνω από 70% με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε οι χώρες που θα συμμετέχουν να υποχρεούνται να μειώσουν το δημόσιο χρέος τους. Ε, αυτό είναι ενισχυτική δημοσιονομική ε, πειθαρχία. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων λένε ότι έτσι θα μειωθούν τα επιτόκια για χώρε όπω η Ιταλία και η Ισπανία για την ανάκαμψη. Σα ρωτάω λοιπόν, γιατί δεν το κάνετε αυτό το πράγμα. Διότι με τρόπο ευφυή e θα μπορούσαμε να λύσουμε βραχυπρόθεσμα την κρίση. Να πω κάτι όμω, κυρία Μέρκελ, το κοινοβούλιο αυτό έχει αποφανθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Διαπραγματευόμαστε, ε, διαπραγματευόμαστε και για τη συμφωνία των δύο σημείων και των έξι προτάσεων του ΣΚΕΣΙΚ ε, ε, και ε, εκεί ε, ακόμη δεν υπάρχει η προβλεπόμενη αυτή λύση που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Κύριο, κύριο Σβόμποντα. Κυρία ε, Καγκελάριε, είπατε ότι είστε φυσικός. Βεβαίως, ε, ε, εμείς τις τις μεταρρυθμίσεις μπορούμε να τις κρίνουμε με διαφορετικό τρόπο. Πάντως ε, είναι τελείως διαφορετική η μεταρρύθμιση που έγινε στη Γερμανία και αυτή που πιέζεται να κάνει η ε, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά ζητούνται άλλα πράγματα επί τόπου, ασκούνται άλλες πιέσεις. Γιατί πέρασαν δύο χρόνια στην Ελλάδα, για παράδειγμα, για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και γιατί καθυστέρησε δύο χρόνια η λίστα Λαγκάρντ. Εκεί πρέπει να δοθούν ε, προτεραιότητες. Η φοροδιαφυγή δεν ε, είναι παραδεκτή και πρέπει να καταπολεμηθεί. Δεν το συζητώ. Κάτι στο οποίο συμφωνούμε. Αυτό που είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο, και εγώ συμφωνώ μαζί σα, ανήκει στην Ευρώπη το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έπρεπε το Ηνωμένο Βασίλειο να μείνει στην Ευρώπη. σω θα έπρεπε να πείτε ε, στον κύριο Κάμπρα να πηγαίνει πιο συχνά στο City του Λονδίνου ε, θα, ε, οι λαϊκιστές, ο κ. Φαράτζ ε, έχουν διαφορετική γνώμη, αλλά νομίζω ε, ότι ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το λαό. Δεν θα πρέπει να, κάνουμε, να κάνουμε κριτική στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συζητήσεις περί εξόδου από την Ευρώπη. Τέλος για τον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε έναν ορθολογικό προπολογισμό και για την ανάπτυξη και για πολλά άλλα. Πολλά μπορείτε να πείτε στον κύριο Κάμερον εδώ, γιατί οι Βρετανοί ήταν υπέρ της διεύρυνσης, έδωσαν μάχη γι' αυτό. Καλώς. Και τώρα λένε ε, οι Βρετανοί, οι Πολωνοί και άλλοι διαβάστε το, την ε, λόγο του Πολωνού ε, Πρωθυπουργού, τώρα ε, λέει, τώρα είστε μέσα, δεν χρειάζεστε άλλα χρήματα από εμά. Όποιο είναι για την διεύρυνση, και εγώ ήμουν πολύ υπέρμαχο τη διεύρυνση, πρέπει όμω να διαθέτουμε σε αυτού που έχουν ανάγκη τα απαραίτητα κονδύλια. Κάθε τι, οτιδήποτε άλλο είναι άδικο. Πρέπει να είναι δίκαιο ο προπολογισμό. Να πείτε στον κύριο Κάμερον ότι εδώ υπάρχει μια ισχυρή βούληση αν υπάρξει βέτο στον προπολογισμό και απορριφθεί και αν υπάρξουν μεγάλες μαζικές περικοπές, τότε θα δώσουμε μάχη ούτω ώστε να υπάρξει ένας ρεαλιστικός προπολογισμό στην Ευρώπη με προσανατολισμό στην ανάπτυξη. Και εμεί μπορούμε να επιδείξουμε πυγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα το κάνουμε ε, αυτή τη φορά, ελπίζοντα την υποστήριξή σα, κυρία Καγκελάρη. Θέλω να υποστηρίξω το φιλικό διαζύγιο του κύριου Φέραντζ, αλλά επιτρέψτε μου ε, να, σας πω, να σας επιστήσω την προσοχή στην κυδαιμονία των 27 παιδιών των άλλων κρατών μελών. Εάν πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε το φιλικό ε, διαζύγιο, πρέπει να συζητήσουμε και για την κυδαιμονία των παιδιών, όχι μόνο των 27 κρατών μερών, αλλά και της Βρετανίας. Κυρία Καγκελάρη, έχετε δίκιο. Πρέπει να δράσουμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αλλά το είπατε δεν θα απαγορεύσουμε στις χώρες που θέλουν να εισέλθουν στο ευρώ, που δεν έχουν εισέλθει ακόμα, να συνεχίσουν να εργάζονται για αυτή την αλληλεγγύη. Πάνω σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πάνω σε αυτή την αλληλεγγύη έχω και μια άλλη πρόταση. Ο ε, αρχηγός του Βρετανικού κράτους, όπως το είπε και ο συνάδελφος, ε, τα βρετανικά χρήματα, όπως το είπε και ο συνάδελφος Σβόμποντα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αλληλεγγύη, αλλά πρέπει ο προπολογισμό να είναι σοβαρός και για να είναι σοβαρός θα πρέπει το 80% ε, των χρημάτων να ξαναγυρνάνε, να επιστρέφουν στις επενδύσεις. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ, κύριε Κάλαναν, δεν ελήφθησαν, ελήφθησαν με πλειοψηφία και ψηφίσαμε με πλειοψηφία εδώ στο, Κοινοβούλιο, οπότε αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Κυρία Μέρκελ, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Η πολιτική έρευνας και καινοτομίας. Είχαμε μεγάλη συζήτηση σήμερα το πρωί στην ομάδα μας. Όλοι μιλούμε για την πολιτική έρευνας και καινοτομίας. Πού είναι, πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία, πού είναι η σχετική πολιτική που πρέπει να στηρίξουμε. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε γρήγορα και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό με εκθέσεις πρωτοβουλίας ούτε μόνο με βάση την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, την απασχόληση. Χρειάζεται εδώ να συζητήσουμε με το Συμβούλιο για να βγούμε γρήγορα από αυτό το αδιέξοδο. Βρισκόμαστε σε μια σοβαρή κρίση, θα βγούμε πολύ γρηγορότερα εάν ε, αγγίξουμε εκεί ακριβώς που πρέπει να αγγίξουμε, αν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Παρακαλώ εσείς κυρία Μέρκελ. Σύντομα σε κάποια λίγα πράγματα να ανταποκριθώ. Κυρία Τσίμερ, όσον αφορά τη νομική βάση του Δημοσιονομικού Συμφώνου, πρώτον, θα θέλαμε αυτό να γινόταν στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συνθήκων. Κάποιοι δεν το ήθελαν. Ήθελαν ως προϋπόθεση να έχουμε και άλλες αλλαγές της συνθήκης όσον αφορά την ρύθμιση των οικονομικών αγορών που δεν συμφωνούσαμε εμείς και άλλοι επίσης. Και γι' αυτό ως σε μια διακυβερνητική συμφωνία που υπήρξε, είπαμε με σαφήνα, μέσα σε πενταετή διάρκεια θέλουμε να ενταχθεί στις ευρωπαϊκές συνθήκες, να μην υπάρξουν νέοι πυλώνες ε, αυτοί υπαρκτοί. Και το Συμβούλιο, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου μας είπε ότι η, η, ο δανεισμός αυτός ως δάνειο είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και καλό θα ήταν σε σχέση με την Ευρώπη να μην κλείσουμε αυτόν τον δρόμο, αυτή την πορεία που πρέπει να καλύψουμε. Την χρειαζόμαστε και τουλάχιστον το δυνατόν πιο γοργά πρέπει να επανενταθεί αυτό στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Κυρία Χάρμς προς εμάς, ξέρω ότι πολλά απαιτήθηκαν από τους Έλληνες δεν θέλω καθόλου αυτό να το παρακάμψουμε ή να το αρνηθούμε. Εκείνοι που είναι πολύ πλούσιοι στην, στην Ελλάδα δεν φορολογήθηκαν. Τα βάρη τα έφεραν εκείνοι οι οποίοι ήταν πραγματικά δεν ε, ζούσαν σε καθεστώς ευημερίας, οι μισθωτικοί συνταξιούχοι δηλαδή. Και γι' αυτό παρακαλώ χάρη της ε, ε, δικαιοσύνης να αναφέρουμε ότι η κρατική διοίκηση είναι υδροκέφαλη. Δεν υπήρξε μεταρρύθμιση όταν ε, έπρεπε να γίνει κάτι και σε σχέση με την Πορτογαλία και σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπήρξαν διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα παρότι η αγοραστική δύναμη δεν είναι η μεγαλύτερη διαφορά και σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που ακολουθούνται για να να ακολουθηθεί η οικονομική ανάπτυξη μέσα στην ίδια την ε, οικονομική κρίση η Λιθουανία, η Λετωνία και η Εστονία έκαναν τεράστιες προσπάθειες και μεταρρυθμίσεις και έχουν σήμερα καλά θετικά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης. Πραγματικά και με τους συναδέφους από κοινού ε, τοποθετούμε και έτσι πρέπει να τα δούμε και σε σχέση με τους ε, Σλοβάκους ε, πρέπει να συζητηθεί για παράδειγμα με τους σοσιαλδημοκράτες εκεί το ε, ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι το ότι εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε νέα κράτη-μέλη που πάρα πολλές θυσίες υποχρεώθηκαν να υποστούν και να αντέξουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και σε σχέση με τον κύριο Φερχόφστα δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω να μην ορκίζεστε. Το ότι μπορούμε να αντιπαρατηθέμεθα δείχνει ότι στην Ευρώπη έχουμε την ίδια τοποθέτηση όπως τα εθνικά μας κοινοβούλια σε σχέση με την εσωτερική πολιτική. Εξαιρετικό αυτό. Ούτε και εκεί συμφωνούμε πάντα όλοι μεταξύ μας. Ε, σε σχέση με τους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες, κύριε Σβόμποντα, πρέπει να ε, δείτε πως ε, τους γνωρίζει η κυρία Μέρκελ, λέει ο, λέει ο πρόεδρος κύριος Σούλτς προς την κυρία Μέρκελ. Γνωρίζει τους Γερμανούς σοσιαδημοκράτες ο κύριος Βόμποντα. Λοιπόν, τέρματα τα αστεία, θα ήθελα να πω τώρα. Πέρα από το ότι για την νομική βάση που απουσιάζει πλήρως, θα έπρεπε τουλάχιστον μια αλλαγή των συνθήκων να γίνει. Στη σημερινή κατάσταση δεν μας βοηθάει αυτό καθόλου κανένα από τα κράτη με τη μεγάλη υπερχρέωση δεν θα είχαν την ευκαιρία να αποσβέσουν τα χρέη τους. Και Αντίθετα θα έπρεπε πρώτα και το έλλειμμα να μειωθεί και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη απάντηση και δεν θα υπήρχε λοιπόν ε, δυνατότητα καμία προοπτική αν δεν εγκρίναμε το Ταμείο Διάσωσης. Όμως έλαβα υπόψη τις παρατηρήσεις σας, ε, τις οποίες σημείωσα και θα ήθελα να δώσω δίκιο στον κύριο Σβόβοντα. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν ένα κράτος το οποίο πάντα ανέφερε τα θέματα της διεύρυνσης Ευρώπης. Και όποιος είναι υπέρ της διεύρυνσης Ευρώπης πρέπει να είναι υπέρ της συνοχής και συνεκτικότητας της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μεγάλη κρίση στην Ευρώπη σε σχέση με το ευρώ. Αλλά θα καταλήξουμε και σε μεγάλη κρίση όλοι οι Ευρωπαίοι αν δεν προχωρήσουμε περαιτέρω στην ανάπτυξη της Ευρώπης και αυτό πραγματικά μπορούσαμε να το κάνουμε σωστά στο παρελθόν με τα ταμεία συνοχής, με, με τα διαθροτικά ταμεία δράσαμε ώστε να σε κάποια σημεία θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα. Μάθαμε τα μαθήματά μας. Με μεγαλύτερη ελαστικότητα πρέπει να δρουν τα ταμεία αυτά σε σχέση με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα για να ενδυναμώσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάθαμε αυτά τα μαθήματα. Η Γερμανία από με τη Γαλλία ήταν εκείνα τα κράτη που πρώτα είναι ότι τώρα θα πρέπει να διεξαχθεί αυτή η σύνοδος κορυφής για τα δημοσιονομικά και να μην περιμένουμε περαιτέρω, να μην σταυρώσουμε τα χέρια μας για το ρόλο της Ευρώπης ε, παγκόσμια, για το, το θέμα του ποιες επενδύσεις θα απαιτηθούν για την Ευρώπη όταν δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί το 2014 και δεν γνωρίζουμε ποιος θα επενδύσει και σε σχέση με τις ευρωχώρες και τις χώρες εκτός ε, ευρωζώνης ε, και σε σχέση και με τη χρηματοδότηση Δηλαδή ένα πολύ αρνητικό μήνυμα θα δίναμε αν ε, δεν προχωρούσαμε τώρα. Και όσον αφορά την πολιτική για την έρευνα, φυσικά είμαι υπέρ αυτή. Και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Έρευνα, το οποίο προγάγαμε. Και πρέπει να καταλήξουμε σε ένα πιο εξυγχρονισμένο προσανατολισμό. Και ταυτόχρονα, όταν έχουμε ε, ετήσια ε, αύξηση κατά μεγάλο ποσοστό για το ίτερ, και δεν θέλω να τερματιστεί το ίτερ, όχι, δεν θέλω να τερματιστεί το ίτερ. Δεν ήταν αυτό το μήνυμα, όχι. Πρέπει όμως ε, να κοιτάξουμε ταυτόχρονα πώς τα κονδύλια θα τα χρησιμοποιούμε με τον βέλτιστο τρόπο για την μέγιστη πρόσθετη αξία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Μέρκελ. Κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ κυρία Καγκελάρια. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας τρεις σύντομες επισημάνσεις. Πρώτα απ' όλα, η ανοιχτή διάσκεψη των Προέδρων είχε σαφώς ε, υψηλότερη συμμετοχή από τους Ευρωβουλευτές από ότι κανονικά οι Ολομέλειές μας στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ας μας προβληματίσει αυτό. Δεύτερο, διαπιστώνω κυρία Μέρκελ, ναι, ναι, σε σχέση με την κατάργηση της ε, Twitter. Ναι, έστω. Το δεύτερο σημείο είναι, διαπιστώνω κυρία Μέρκελ και θέλω αυτό ρητά ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευγνωμοσύνη να το λάβω υπόψη από πλευρά σας. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Όλα όσα συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για σας ως σημαντικό μέλος του Συμβουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο εταίρος και ο νομιμοποιητής των πραγμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για αυτήν την τοποθέτηση. Θα ευχόμουν να ήταν αυτό η ομόθυμη, ομόφωνη τοποθέτηση του Συμβουλίου. Έχετε μεγάλη επιρροή. Παρακαλώ ενθαρρύνετε το Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί. Θα ήθελα το εξής να αναφέρω. Πιο πριν αναφέρατε την Λετωνία ο Πρωθυπουργό των εδώ σε αυτή την αίθουσα απίφθινε λόγο προ την κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ. Ο κύριο Ντομπρόφσκη, σε αυτόν τον λόγο που εξεφώνησε ανάφερε τα τεράστια, τις τεράστιες θυσίες που έκαναν οι πολίτε τη χώρα του για να μπορέσουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε αν η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο λαό μου μετά από όλε αυτέ τι θυσίε που υποστήκαμε θα είναι να διαγραφεί, να περικοπεί ο προπολογισμό ώστε να μην διατίθενται πλέον κονδύλια σύνοχή τότε θα γίνει το ίδιο με μάσα όπως ε, η μοίρα του Φίτσο στην ε, ε, Σλοβακία. Δηλαδή θα τερματιστεί η δική μας θητεία, θα είναι το τέρμα πλέον της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πολίτες. Γι' αυτό δεν πρέπει να πάψει η αλληλεγγύη. Ευχαριστώ για αυτό το οποίο αναφέρατε. Στο τέλος για τους ε, Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες ε, είπατε πρώτον σε εμά είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την Ομοσπονδιακή Βουλή και δεύτερον οι σοσιαλδημοκράτες είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή πολιτική. Νομίζω αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Σας ευχαριστώ.